Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann eröffne ich die Sitzung des Handelsausschusses. Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Καλώς ορίσατε όλοι μετά τις θερινές διακοπές. Ελπίζω να περάσατε καλά και να είσαστε πλέον ξεκούραστοι και να ήρθατε να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις των επόμενων εβδομάδων στον τομέα του διεθνούς ε, εμπορίου, που είναι και το μέσα αρμοδιότητα της Επιτροπής μας, έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε. Και έτσι περνάμε λοιπόν στην ημερήσια διάταξη, στο σημείο 1. Δεν ξέρω αν υπάρχουν οποιαδήποτε επιθυμίες να αλλάξει η ημερήσια διάταξη. Όχι. Μάλιστα λοιπόν έτσι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Στο 2 της ημερήσιας διάταξης ε, έγκριση των πρακτικών της τελευταίας συνεδρίασης της 22ης Ιουλίου. Ο κανόνας είναι και ισχύει πάντα ότι αν μέχρι τα τέλη της συνεδρίασης δεν υποβληθούν ενστάσεις, θεωρείται ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Ωραία. Αυτή λοιπόν την ε, διαδικασία θα ακολουθήσουμε στο 3 του, της σημερινής διάταξης έχουμε τις ανακοινώσει του Προέδρου. Καταρχάς θα ήθελα να σας επενθυμίσω ότι η συνεδρίαση θα μεταφέρεται, μεταβάζεται στο διαδίκτυο. Κατά δεύτερον, σας διαβιβάσαμε τα σχετικά έγγραφα που μπορείτε να δείτε ποιες επιστολές έχουν καταρτιστεί και αποσταλεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις εμπορικέ εξελίξεις, να σας κάνω κάποιες ε, ε, μικρές ανακοινώσεις. Καταρχάς θα ακούσατε ότι οι εξελίξεις μετά το Μπαλί ήταν μάλλον αποθαρρυντικές σε ό,τι αφορά το Trade Facility Agreement, αυτή την ε, συμφωνία για την ευκόλυνση του εμπορίου άρθηκαν φραγμοί λόγω των δραστηριοτήτων της Ινδίας και το Δημόσιο Φόρουμ ε, του ΠΟΕ θα είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε προκειμένου να δώσουμε μια καινούργια όθηση στις συζητήσεις. Για το εμπόριο σε ό,τι αφορά και τις ρωσικές αντιδράσεις, τις ε, κυρώσεις, ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά την απαγόρευση εισαγωγών τροφίμων από τη Ρωσία. Θα πρέπει να δούμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στους Ευρωπαίους παραγωγούς και να προσπαθήσουμε να τις απαλύνουμε. Ο προσκεκλημένος μας θα τα αναλύσει αυτά, αλλά ο, το Συμβούλιο υποστήριξε τα μέτρα που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έτσι θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να εξετάζει ε, προσεκτικά τις επιπτώσεις ε, των κυρώσεων αυτών, των απαγορεύσεων αυτών στους Ευρωπαίους παραγωγούς και μετά θα προτείνει και αντίστοιχα μέτρα απάλληλης του φαινομένου. Ύστερα, συνάδελφοι, στι δύο τελευταίε συνεδριάσει ελήφθησαν περαιτέρω αποφάσει σε ό,τι αφορά τα EPA, σε ό,τι αφορά την ε, Νότια Αφρική. Άρα στο μέλλον θα κληθούμε να εξετάσουμε και τα θέματα αυτά σε ό,τι αφορά το EPA, τη Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης, δηλαδή με το Καμερούν. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, κάτι άλλο σε σχέση με τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ό,τι αφορά τις ε, διαπραγματεύσεις teaser. Δημοσιεύτηκαν σχετικά έγγραφα από ευρωπαϊκής πλευράς και νομίζω ότι σωστό είναι στο πλαίσιο αυτό και των ε, σχετικών διαβουλεύσεων να υπάρχουν ε, αντικειμενικά, επιστημονικά στοιχεία, προκειμένου η κοινωνία των πολιτών να έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί σωστά το τι αποτελεί το αντικείμενο διαβουλεύσεων. Και θα δημοσιευθούν τα σχετικά έγγραφα. Τελευταία ανακοίνωση τώρα στην άνταλφη θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της Ουκρανίας και της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης. Θα γνωρίζετε ότι η Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης, η οποία επί της ουσίας πραγματεύεται εμπορικά ζητήματα, αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την σταθεροποίηση της οικονομικής κατάστασης στην Ουκρανία. Και σε μια κοινή δήλωση του Προέδρου της ε, Επιτροπής και ε, μου, αποφασίσαμε ότι θέλουμε το συντομότερο δυνατόν να ψηφίσουμε αυτή την ε, συμφωνία με την Ουκρανία και έτσι κατακτήσαμε ένα πολύ αυστηρό χρονοδιάγραμμα. Ωστόσο, εκ των υστέρων αποδείχθηκε ότι αυτό το χρονοδιάγραμμα πρέπει να γίνει ακόμα πιο αυστηρό, να διαμορφωθεί ακόμα πιο αυστηρά, γιατί η επικύρωση από, το, α, επικύρωση από την Ουκρανία, από πλευρά Ουκρανία, πρέπει να γίνει από το τρέχον κοινοβούλιο. Το Οκτώβριο, ξέρετε ότι έχουμε εκλογέ στην ε, Ουκρανία. Και έτσι λοιπόν ε, έγιναν συζητήσει μεταξύ του Προέδρου τη Ουκρανία και του, του, του Προέδρου του Κοινοβουλίου μα το Σαββατοκύριακο που μα πέρασε, προκειμένου να συμφωνηθούν τα σχετικά και έτσι εκφράστηκε λοιπόν η επιθυμία και συμφωνήθηκε ότι η επικύρωση της ε, συμφωνίας εταιρική σχέσης θα πρέπει παράλληλα ουσιαστικά να εγκριθεί στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η εβδομάδα λοιπόν της, 10... της 5ης έως 18ης Σεπτεμβρίου. Ε, Σεπτεμβρίου συγγνώμη. Ε, δηλαδή η επόμενη εβδομάδα της Ολομέλειας στο Στρασβούργο. Πιστεύω ότι δεδομένη της κατάσταση, η οποία είναι ασφαλώς ιδιαίτερο ε, έκτακτη, αυτό το βήμα τη παράλληλης επικύρωσης στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι αρκετά λογικό. εξαίρεση. Και μάλιστα κατεξαίρεση ε, επιτακτικό αυτό το μέτρο. Αυτό που σημαίνει ότι εμεί ως Επιτροπή ε, δεν θα είμαστε σε θέση να γνωμοδοτήσουμε για τη συμφωνία αυτή λόγω των χρονικών περιορισμών. Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων την επόμενη εβδομάδα θα κάνει μια έκτακτη συνεδρίαση προκειμένου να καταρτήσει τις συστάσεις από πλευρά της Επιτροπής για την Ολομέλεια και έτσι στις 15, από τις 15 Σεπτεμβρίου και μετά να μπορεί να ψηφιστεί το κείμενο από την Ολομέλεια. Δεν μπορεί λοιπόν να αντιεξαχθεί η διαβίλευση η οποία θα κατέληγε ενδεχομένω σε γνωμοδότηση. Θα καταλαβαίνετε ασφαλώς ότι ως πρόεδρος της Επιτροπής δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένο για το αυστηρό αυτόχρονο διάγραμμα που δεν μας επιτρέπει να καταρτήσουμε γνωμοδότηση. Αλλά δεδομένη της πολιτικής κατάστασης και της πολιτικής ανάγκης θεωρώ ότι θα πρέπει κατ' εξαίρεση να αποδεχτούμε την κατάσταση αυτή. και να μην ξεκινήσουμε θεσμικούς αγώνες και θεσμικές μάχες για το θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά, θα αποστείλουμε μία επιστολή στην ΑΦΕΤ, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, με τη σαφή διευκρίνηση ότι η κατάσταση αυτή είναι σαφώς ε, ασυνήθιστη. Αποτελεί εξαίρεση και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προηγούμενο για μελλοντικέ περιπτώσεις. και να μεταβιβάσουμε, να διαβιβάσουμε κάποιες παρατηρήσεις προς την Επιτροπή ΑΦΕΤ σε ό,τι αφορά τα θέματα περιεχομένου. Το θέμα αυτό θα το εξετάσουμε και λίγο πιο επισταμένος σήμερα το απόγευμα, αλλά εν πάση περιπτώσει ήθελα να το θίξω. Δεν ήθελα να ξεκινήσω συζήτηση για τα θέματα αυτά, γιατί θα, θα έχουμε την ευκαιρία αυτή και σήμερα το απόγευμα. Αλλά στο επόμενο σημείο της ημερής της διάταξης έχουμε έναν προσκεκλημένο και νομίζω ότι κάποια από τα θέματα αυτά θα μπορέσουμε να τα συζητήσουμε και με τον προσκεκλημένο μας. Θα ήθελα λοιπόν να περάσω στο επόμενο σημείο της της διάταξης, το 4 δηλαδή, γλωσσικό προφίλ στην Επιτροπή μας. Πρέπει να διατίθεται κάθε επίσημη γλώσσα. Αλλά από την άλλη καλούμαστε να δημορφώσουμε και ένα αποτελεσματικό, αποδοτικό γλωσσικό προφίλ. Δηλαδή δεν έχει νόημα να παρέχετε μια γλώσσα που, για την οποία δεν υπάρχει βουλευτής. Άρα λοιπόν το γλωσσικό προφίλ διαμορφώνεται ως εξή. Και επειδή η αίθουσα έχει και 16 καμπίνες, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, ολλανδικά, ελληνικά, μπορείτε και να ακούτε και να μιλάτε, τσαχικά, πολωνικά, ρουμάνικα, ισπανικά, πορτογαλικά. στις 12 καμπίνες όπως, ε, σε αίθουσα με 12 καμπίνες όπως η αίθουσα αυτή. Οι γλώσσες είναι γερμανικά, αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ολλανδικά. Ελληνικά σε κάθε περίπτωση μπορείτε να μιλάτε και να ακούτε. Καλημέρα σας. Αν ε, θέλετε κάτι διαφορετικό, φυσικά θα το σημειώσουμε. Θα το λάβει υπόψη ασφαλώς η γραμματεία, σε περίπτωση που υπάρχει επιθυμία για κάποια άλλη γλώσσα, προκειμένου κανένας συνάδελφος να μην αισθάνεται ε, ότι μειονεκτεί. Αν μέχρι τέλος της συνεδρίασης δεν υπάρξει οποιαδήποτε ένσταση, θα ακολουθήσουμε λοιπόν το καθεστώς αυτό. Ωραία, περνάμε λοιπόν τώρα στο προσκεκλημένο μας. Buongiorno. Καλημέρα σας και χαίρομαι ιδιαίτερος που έχουμε μαζί μας σήμερα τον Κάρλο Καλέντα, τον Υφυπουργό Εμπορίου και Οικονομικών Εξελίξεων της Ιταλίας. προκειμένου να μας παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Ιταλικής Προεδρίας. δεδομένων και των εκλογών και των διάφορων διαδικασιών που έπρεπε να ακολουθήσει το Κοινοβούλιο. Δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ιδιαίτερα με την Προεδρία. Γι' αυτό λοιπόν είναι ιδιαίτερα σημαντική αυτή η συνάντηση και νομίζω ότι έχουμε κάποια πολύ σημαντικά στοιχεία στην ε, διάταξη για σήμερα. Να τα θέσουμε, τα Trade Defense Instruments, τα εργαλεία, τα μέσα υπεράσπιση του εμπορίου και πολλά άλλα, τα οποία θα δείξουμε. Οι διαπραγματεύσεις για εμπορικά θέματα. Ενδεκτικά αναφέρω τα θέματα αυτά και θα ήθελα να δώσω πάρα αυτά λοιπόν το λόγο στον Υφυπουργό. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκεται μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Μέλη της Επιτροπής. Είναι τιμή για μένα να έχω την ευκαιρία να μιλήσω μπροστά στην Επιτροπή σας για να παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Ιταλικής Προεδρίας σε θέματα εμπορικής πολιτικής. Βρισκόμαστε στην αρχή της θητείας και πιστεύω ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσει μια συζήτηση για το στρατηγικό ορίζοντα εντός του οποίου θα πρέπει να λειτουργήσουμε τα ερχόμενα χρόνια. Οι επιλογές της εμπορικής μας πολιτικής τις οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα επόμενα χρόνια θα είναι πλέον σημαντικές εδώ και πολύ καιρό για αυτή την περιοχή του κόσμου. Βρισκόμαστε ε, στην έναρξη μια νέα φάση τη παγκοσμιοποίηση και εμεί στην Ευρώπη θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να είμαστε πρωταγωνιστέ ή να ε, υποστούμε την ενεργό δράση άλλων μεγάλων πρωταγωνιστών στο παγκόσμιο προσκήνιο. Δεν υπάρχει τρίτη εναλλακτική. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον περασμένο Ιούνιο καθόρισε μια νέα ατζέντα για την ανάπτυξη και την απασχόληση που ονομάστηκε Στρατηγική Ατζέντα για την Στρατηγική Ένωση σε καιρού αλλαγή. Το αξίωμα αυτή τη πορεία είναι ότι όλε οι πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμβάλλουν στο να επιτύχουμε του ε, σκοπού και του στόχου τη ανάπτυξη, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Αυτό ισχύει περισσότερο για την εμπορική πολιτική, η οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη τι ιδιαιτερότητε αυτή τη χρονική φάση που περνά η παγκόσμια οικονομία και το νέο τη νέα φάση που περνάει παγκοσμιοποίηση. Θα ήθελα εδώ να τονίσω τρεις ε, πτυχές αυτής της νέας φάσης της παγκοσμιοποίησης, αν θέλουμε να εκπονήσουμε μια αποτελεσματική στρατηγική. Πρώτα απ' όλα η διαφορά στο κόστος παραγωγής μεταξύ των ε, προηγμένων και των λιγότερων προηγμένων χωρών ουσιαστικά ε, γίνονται ολοένα και μικρότερες. Έχουμε μια, ένα φαινόμενο Μετατόπιση των επιχειρήσεων που πιστεύω ότι θα επιτυχηθεί τα ερχόμενα χρόνια. Θα μπορέσουμε να αποφεληθούμε από αυτό το φαινόμενο που έχει ονομαστεί και reshoring μόνο αν είμαστε σε θέση να έχουμε μεγαλύτερη δραστηριότητα επιχειρηματική στην Ευρώπη. Με λίγα λόγια, θα πρέπει να υπάρξει μια κίνηση προ τη Δύση. Αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι η Ευρώπη θα συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία αν δεν λάβουμε μέτρα. Επίση, οι αναδυόμενε οικονομίε έχουν τάσει προστατευτικέ, ιδίω με τον υπόγειο τρόπο των μη δασμολογικών φραγμών. Αυτό το φαινόμενο δεν αφορά μόνο τις χώρες που έχουν ε, πρόσφατα εκβιομηχανιστεί. Θα πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε ότι ένας ε, κόσμος που έχει γίνει ενιαίος στην ουσία διαιρείται παρόλα αυτά μεταξύ χωρών που έχουν αποδεχτεί τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς και αυτές που έχουν νεοπροστατευτικές τάσεις. Οι συμφωνίες για τις ελεύθερες συναλλαγές ε, που είναι διμερούς χαρακτήρα και βασίζονται στο πολυμερέ σύστημα, είναι μία πρώτη τάση, μια πρώτη απόδειξη αυτής της νέας τάσης. Επίσης, για να έχουμε ε, πραγματικά προϊόντα κατασκευαστικά και ε, για να ικανοποιήσουμε την παγκόσμια ζήτηση, θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ικανοποιούμε και τις διαφορετικές ανάγκες που απαιτούν οι συναλλαγές σε ένα παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο. Θα ήθελα να ε, πετύχουμε ένα 20% παραγωγής του ένα 20% του ΑΕΠ για την παραγωγή τέτοιων προϊόντων μέχρι το 2020. Αυτός ο στόχος ε, θα καθοριστεί βεβαίως από το τι εμπορική πολιτική θα προβλέψουμε και εξαρτάται και από τον παραγωγικό μας ιστό, δηλαδή από την απασχόληση αλλά και από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι βασικά συμπληρώματα με τις δεξιότητες και την καινοτομία που μπορούν να παρουσιάσουν για τις μεγαλύτερε επιχειρήσει μας. Στο επίκεντρο αυτής της ε, στρατηγικής για την εμπορική μας πολιτική τα ερχόμενα χρόνια θα χρειαστεί να έχουμε και νέες ε, συμφωνίε και τις ελεύθερες συναλλαγέ με ε, μια επίτευξη ολοένα και πιο βραδία αλλά σε πολυμερές επίπεδο οπωσδήποτε. Το νέο σύστημα συναλλαγών νομίζω θα παρουσιάσει πλέον τρία επίπεδα, όπου οι διμερείς συμφωνίες θα είναι η εμπροστοφυλακή της παγκοσμιοποίησης, ενώ οι πολυμερείς συμφωνίες για τα πράσινα αγαθά λόγου για τις υπηρεσίες ε, πληροφορίας και τεχνολογίας, θα ε, επιτυχάνονται σε τομεακή βάση για τις χώρες που ενδιαφέρονται για του είδους ε, συναλλαγών. Και βεβαίως το ίδιο και για τις ε, συμφωνίες που θα επιτυγχάνονται στα πλαίσια το, της Ντόχα και της σχετικής ανάπτυξης, ατζέντα ανάπτυξης. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να συνεργαστούμε και να είμαστε θετικοί με όλες τις χώρες ε, και να μην έχουμε ιδεολογικές προσεγγίσεις από τα θέματα προκειμένου να γίνει καθοριστική ε, η βασική πορεία της εμπορικής μας πολιτικής η επίτευξη τέτοιων συναλλαγών. Με την επιτυχία των διαπραγματεύσεων στον Παλί που είδαμε ότι μερικές χώρες δεν ακολούθησαν ιδιαίτερα υπεύθυνη στάση, θα πρέπει εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες που έχουν την ίδια, ε, το ίδιο σκεπτικό με εμά να προχωρήσουμε σε αυτό το δρόμο και κάποιες χώρες να αποδεχθούν τις αναπόφευκτες ε, επιλογές που θα πρέπει να κάνουν. Δεν είναι καθόλου εύκολο για κανένα σε αυτή τη φάση να μείνει στο περιθώριο. Επιτρέψτε μου να σταθώ εδώ στη συμφωνία με τον Καναδά. Η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ήταν λόγος ικανοποίηση για όλους. Θα πρέπει να ε, μπορέσουμε εδώ να φέρουμε εις πέρας αυτή τη συμφωνία και να την υλοποιήσουμε με ικανοποιητικό τρόπο. Ε, έχουμε θετικά αποτελέσματα από τη συμφωνία αυτή για όλους τους τομείς που αποσχολούν την εμπόρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως για τους δασμούς. Οι δημόσιες προμήθειες είναι πλέον ε, απελευθερωμένες και υπάρχει μια πιστική συμφωνία ότι θα αναγνωριστούν οι γεωγραφικές ενδείξεις που είναι πολύ σημαντική για την εξαγωγή ε, γεωργικών προϊόντων. Γενικότερα πρόκειται για μια συμφωνία που θα αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς κάτι που θα είναι ένα πεδίο ε, που θα έχουμε εξερευνήσει για τις σημαντικότατες διαπραγματεύσεις που θα έχουμε το επόμενο διάστημα, τις συμφωνίες με τις, την, διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα, ε, χρειάστηκαν 7 χρόνια για να επιτύχουμε την συνολική οικονομική και εμπορική συμφωνία. Δεν μπορούμε λοιπόν να καθυστερήσουμε το ίδιο για τι διαπραγματεύσει TTIP. Είναι η πλέον σημαντική συμφωνία που θα έχουμε διαπραγματευτεί ποτέ με τον πλέον ε, σημαντικό εμπορικό μα εταίρο. Και αυτό στη νέα καμπή που έχει λάβει παγκοσμιοποίηση. Για το θέμα του TTIP ε, έχουμε ακούσει πολλά διαφορετικά νέα και απόψει. Υπάρχουν πολύ μεγάλε τάσει όπιστο και επίσης ε, πολλές, ε, πολλοί μύθοι και πολλές φήμες σε σχέση με τον απόρριτο χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων. Υπάρχουν βεβαίω κάποιε τυπικέ προποθέσει που πρέπει να γίνουν σεβαστέ, αλλά θα πρέπει σε συνεργασία με τον Επίτροπο του Εμπορίου ε, την επιστολή που αποστήλαμε στο Συμβούλιο να την συνυπογράψουμε για να υπάρξει ουσιαστικά διαφάνεια στην διαπραγματευτική εντολή και να γίνει μια μεγαλύτερη προσπάθεια για σαφήνεια και διαφάνεια ακριβά, για, ε, ακριβώς, για να δούμε ακριβώς τα θέματα που διακυβεύονται εδώ. Με την ε, δημοσιοποίηση αυτή των διαπραγματεύσεων θα καταλάβουμε ποια ακριβώς θέματα έχουν συμπεριληφθεί στις διαπραγματεύσεις και ποια όχι και ποια ακριβώς ενδιαφέρουν το κάθε κράτος μέλος. Έτσι θα πρέπει να παρακολουθούμε στενά το πώ εξελίσσεται το κάθε γύρο των διαπραγματεύσεων. Αλλά κάτι που θα πρέπει να έχουμε ευθύ εξ αρχή σαφέ στο μυαλό μα είναι ότι οι διαπραγματεύσει TTIP θα πρέπει καταρχά να ωφελήσουν τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Δεν είναι μία ε, συμφωνία που σκοπό έχει να ευνοήσει τι ε, πολυεθνικέ. Αυτό είναι πραγματικά παραπλανητικό. Οι πολυεθνικέ εταιρείε ήδη λειτουργούν πέρα από τα σύνορα και μπορούν να ε, καλύψουν τη ζήτηση εκεί που την εντοπίζουν. Η μη δεσμολογική φραγμή και η ε, ρυθμιστική ευθυγράμμιση θα ε, ευνοήσουν κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εκείνες που δεν έχουν τους πόρους για να αντιμετωπίσουν εμπόδια και γραφειοτικούς φραγμούς στις διάφορες οικονομίες. Κατά τον ίδιο τρόπο είναι σαφές ότι τα συστήματα πρόνοιας και από τις δύο ε, όχθες του Ατλαντικού δεν θα πρέπει να πληγούν από αυτή τη συμφωνία, καθώς εκτός των διαπραγματεύσεων θα παραμένουν και κάποια θέματα που θα έχουν να κάνουν με διατροφική ασφάλεια και τις πολιτιστικές διαφορές. Ε, οπωσδήποτε η περίπλοκες, τα περίπλοκα ζητήματα που αφορούν αυτέ τι διαρματεύσει είναι πολλά και θα πρέπει να εμβαθύνουμε σε αυτά. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εντείνει τι προσπάθειε τη σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Χρειάζεται εδώ συλλογική εργασία και ο δικό σα ε, πολύτιμο ρόλο, ε, καθώ είσαστε οι άμεσοι εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών λαών. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στα πραγματικά ζητήματα τη ουσία και όχι αυτά που προκύπτουν από ιδεολογικέ προκαταλήψει ή από, έναν, ε, από τις τάσει, που κάποιε φορέ είναι ακατανόητε σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε. Σίγουρα υπάρχουν διαφορέ μεταξύ Ευρώπη και Αμερική και πολλέ φορέ είναι και ε, επί τη ουσία, Λόγου χάρη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αποτιμήσει με πολλού διαφορετικού τρόπου το αποτέλεσμα των ε, διαπραγματεύσεων, των δημόσιων διαβουλεύσεων μάλλον και το μηχανισμό ISDS που θα καθορίσει το πώς θα εξελιχθούν οι επενδύσεις με τρόπο που να είναι πιστικός για όλα τα κράτη-μέλη. Κανείς δεν θα μπορεί λοιπόν, εφόσον ολοκληρωθούν και αυτές οι διαβουλεύσεις, να αποφύγει τις ευθύνε του. Αυτά όμως που μας χωρίζουν από τις ΗΠΑ είναι λιγότερα από αυτά που μας ενώνουν μαζί τους. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή τη δεύτερη χρονική φάση της παγκοσμιοποίησης. Θα πρέπει να ε, εντείνουμε το ρυθμό των διαπραγματεύσεων που μέχρι τώρα ήταν ικανοποιητικό. Είναι πολύ σημαντικό να παρουσιάσουμε και δημοσίω τη σημασία των διαπραγματεύσεων TTIP, γιατί θα υπάρξουν θα υπάρξει πραγματικό αντίκτυπο στι οικονομίε όλων των κρατών μελών. Βεβαίω, η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων αυτών ε, τοποθετείται σε ένα μακρινό ορίζοντα. Περιμένουμε όμω ήδη την ολοκλήρωση του επόμενου γύρου των διαπραγματεύσεων και ελπίζουμε να ολοκληρωθεί η συμφωνία έως έω το τέλο του 2015. Το Συμβούλιο των Υπουργών τον Οκτώβριο θα συζητήσει τα αποτελέσματα του πολιτικού stock taking, όπω ονομάστηκε, ε, των πρώτων δηλαδή αποτελεσμάτων, ε, από τι αρχέ του φθινοπόρου και θα οργανωθούν και δημόσιε ε, με, συμμετοχή του Αμερικανού διαπραγματευτή Μάικ Φρόμαν. Εδώ λοιπόν θα πρέπει εν ώψη του πρόοδου που θέλουμε να επιτελούμε πολύ καλά την στρατηγική που ακολουθούμε στις διαπραγματεύσεις. Να δούμε ότι υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες σε κάποια κεφάλαια των διαπραγματεύσεων που παραμένουν, αλλά ίσως δεν είναι επί της ουσίας και να τα ξεπεράσουμε αυτά για να προχωρήσουμε αλλά και η πορεία των διαπραγματεύσεων θα επηρεάσει και το επηρεάζεται από το πολιτικό χρονοδιάγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών με τις διάμεσες εκλογές της θητείας στο 2015 και βεβαίως τις ερχόμενες προεδρικές εκλογές. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Επ' αυτού λοιπόν θεωρούμε ε, ως Ιταλική Προεδρία ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές δεν θα πρέπει να επιβραδυνθεί ο ρυθμός των διαπραγματεύσεων και ότι μπορούμε να ελπίζουμε σε μια ενδιάμεση συμφωνία εντός του 2015 επί των ουσιαστικότερων ε, κεφαλαίων των διαπραγματεύσεων και εκεί που υπάρχουν λιγότερες διαφωνίες. Και μετά για τα υπόλοιπα θέματα μπορούμε να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις. Ως Προεδρία θα θέλαμε να υπάρχει μια... Ε, πολύ συνετή συζήτηση και πολύ καλά διαφρομένη ε, τόσο επίπεδο του Συμβουλίου αλλά και με την ε, συμβολή του Ευρωκοινοβουλίου. Τώρα, για τι υπόλοιπε διαπραγματεύσει που μα ε, απασχολούν αυτόν τον καιρό, θα περάσω σε μια άλλη χώρα, ο ΑΣΕ, την Ιαπωνία, που είναι και αυτή στρατηγικό μα εταίρο. Είναι γνωστή η σημασία τη Ιαπωνική Αγορά για το διεθνέ εμπόριο και το τι ωφέλη μπορεί να προκύψουν από την ευρωπαϊκή αγορά με μια τέτοια συμφωνία. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη μα τα επιθετικά και αμυντικά δικαιώματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. το πώ μπορεί να υπάρξει απαλληφή των ε, δασμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση και άρση των μη δεσμολογικών φραγμών από την πλευρά της Ιαπωνίας, κάτι που προβλέπεται μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Ήδη τον Ιούνιο είχαμε ένα πρώτο γύρο με τη ρήτρα ραντεβού όπως ονομάστηκε, για να μπορέσουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων. Ε, πολλά τα επίπεδα σε αυτή τη νέα καμπή της παγκοσμιοποίησης, εφόσον θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο χώρο ελεύθερων συναλλαγών που θα μπορεί να προκύψει από την παράλληλη επίτευξη πολλών συμφωνιών από αυτές που συζητούνται η συμφωνία TTIP παραλληλίζεται με τη συμφωνία που αφορά τις ε, σχέσεις στην περιοχή του Ειρηνικού, τις οποίες δημοκρατεύονται οι Ηνωμένε Πολιτείε. Εκεί θα μπορούσε να δημιουργηθεί με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια περιοχή συναλλαγών που θα αφορά το 60% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Μια τεράστια ευκαιρία για όλες τις χώρες που ε, κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή να επιστρέψουν στον προστατευτισμό. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να προαχθούν και οι συζητήσεις Ευρώπης με πολλές από τις χώρες ΑΖΕΑΝ, όπως η Σιγκαπούρη, που είναι σημαντικός εμπορικός μας εταίρος ε, μεταξύ των χωρών ΑΖΕΑΝ. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει τις συζητήσεις για τις επενδύσεις. Ε, ακόμη δεν έχει επιληθεί βέβαια το θέμα της διαχείρισης και προστασίας των επενδύσεων για εμπορικά και βιομηχανικά θέματα. Εκεί περιμένουμε τις εσωτερικές διαπραγματεύσεις της Σιγκαπούρης να ολοκληρωθούν για να προχωρήσουμε. Παρακολουθούμε επίσης τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με άλλες χώρες αυτής της περιοχής της Ασίας, κυρίως με το Βιετνάμ. Για την Ταϊλάνδη, οι εξελίξεις των διαπραγματεύσεων ε, σε σχετίζονται βεβαίως και με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις της χώρας αυτής. Η χρονιά που τελείωσε ε, χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερως από τις εξελίξεις στις δημοτεύσεις με την Κίνα όπου είδαμε ότι η Ευρώπη δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά ιδίως ό,τι αφορά τα φωτοβολταϊκά εκεί οι εσωτερικές μας διαφωνίες ουσιαστικά αποδυνάμωσαν την πολιτική της Ένωσης στις σχέσεις με μερικούς από τους ε, σημαντικότερους εμπορικούς μας εταίρους αλλά που είναι και από τους δυσκολότερους θα πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε λίγο πορεία ε, εκπονώντας μια στρατηγική που μακροπρόθεσμα να επιτρέψει την επιτάξη σε των διαπραγματεύσεων σε θέματα επενδύσεων με προοπτική να ολοκληρωθεί μια συμφωνία που θα δημιουργεί έναν ίσο, ένα, ίσους κανόνες ε, συμμετοχής για την κινέζικη αγορά. Θα πρέπει να φροντίσουμε σε πολλούς τομείς ε, να μην ε, ε, να μην συνεχιστεί η διαρθρωτική υποπαραγωγή της ε, κινέζικης οικονομίας γιατί εδώ μπορεί να υπάρξουν στρεβλώσεις στις εμπορικές μας σχέσεις. Θα πρέπει να δράσουμε προληπτικά και με την επίτευξη λύσεων θα μπορούσαμε να ε, επιδιώξουμε να βρεθούν λύσεις που να έχουν μακροπρόθεσμα αποτέλεσμα. Η Ιταλική Προεδρία σε σχέση με την Κίνα ελπίζει να υπάρξει ε, ολοκλήρωση ε, των διαπραγματεύσεων, τομεακών μάλλον διαπραγματεύσεων για τις γεωγραφικές ενδείξεις, ώστε να δείξουμε πόσο ενεργεί είναι η δράση μας για την προάσπιση των ε, παραδοσιακών ευρωπαϊκών προϊόντων. Άλλες διαπραγματεύσεις που είχαν περάσει σε τέλμα εδώ και καιρό, αλλά τώρα ε, μπορεί να επιταχυνθούν, είναι οι διαπραγματεύσει μας με τι χώρε ε, του Συμβουλίου Συνεργασία του ε, Κόλπου. Η χώρες αυτές, με τις χώρες αυτές συζητούμε το θέμα των εξαγωγικών δασμών και η Ιταλική Προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη σημασία και στις διαπραγματεύσεις με την νότια όχθη της Μεσογείου. Εδώ προχωρούν οι διαπραγματεύσεις μας με το Μαρόκο και στο τέλος του Σεπτεμβρίου συνεχίζεται, θα οργανωθεί η υπουργική συνάντηση στις Βρυξέλλες με εκπροσώπηση από υπουργού των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μεσογείου. Βεβαίως οι χώρες ε, της Ανατολικής Γειτονίας είναι κάτι στο οποίο θα δώσει ιδιαίτερη σημασία Γαλλική Προεδρία. Ιδιαιτέρω, διότι θα θέλαμε να προχωρήσουν οι συμφωνίε ελεύθερων συναλλαγών με τη Μολδοβία, τη Γεωργία και την Ουκρανία. Για την τελευταία αυτή χώρα, κανεί δεν παραβλέπει τη στατική σημασία που έχει εμπορική πολιτική σε αυτήν την ευαίσθητη περίοδο και πόσο αυτή ε, ε, εμπλέκεται ακριβώ με τι πολιτικέ και εμπορικέ προτεραιότητε τη Ρωσική Ομοσπονδία. Εδώ η ασφάλεια στην Ευρώπη, ε, όπως ε, θα την, σχεδιάσουμε για το μέλλον, σχετίζεται και με την ε, δημοκρατία και τις δικές μας αξίες, όπως τις ανταλαμβανόμαστε. Σίγουρα η εμπορική πολιτική μας αντικατοπτρίζει, θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τα συμφέροντά μας στον τομέα της οικονομίας, αλλά η εξωτερική μας πολιτική θα πρέπει να αντικατοπτρίζει και εκείνη και τα συμφέροντα και τις αξίες μας. Η Ιταλία δίνει μεγάλη σημασία στις εξωτερικές μας προς τη Ρωσία, αλλά πρέπει πάντοτε να έχουμε υπόψη και τις προτεραιότητες της εξωτερικής μας πολιτικής. Γι' αυτό θα παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή τις εξελίξεις στις εμπορικές σχέσεις, προκειμένου να μην δημιουργήσουν γενικότερα πολιτικά προβλήματα. Θα παραμείνει ανοιχτό, ανοιχτός ο διάβλος του τεχνοκρατικού διαλόγου μας, προκειμένου να αποφύγουμε εμπορικές στρεβλώσεις και βλέπουμε τα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνει η ρωσική πλευρά. Γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε να μην υπάρξει ε, η υποκατάσταση των ε, εισαγωγών και Γι' αυτό η Ιταλική Προεδρία πρόσφατα εργάστηκε τι τελευταίε εβδομάδε για να αντιμετωπίσει αυτόν τον αρνητικό αντίκτυπο που κινδυνεύει να δημιουργηθεί. Όσο για τη Λατινική Αμερική, ε, θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσει μα με τι χώρε Μερκοσούρ, προκειμένου να επιταχυνθεί η υποβολή ε, προσφορών από τι χώρε αυτέ. Συνεργαζόμαστε στενά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ αυτό το σκοπό. Και ήδη ολοκληρώσαμε πρόσφατα τις ε, συμφωνίε εμπορικών συναλλαγών με το Εκουαδόρ και την Κολομβία. Θα πρέπει λοιπόν από κοινού να δεσμευτούμε για να στηρίξουμε τον πολυμερή διάλογο σε επίπεδο ΠΟΕ. Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου παραμένει η βασική πλατφόρμα όπου μπορούμε ε, να κάνουμε βήματα πρόοδου ουσιαστικά για να προχωρήσουν ταυτόχρονα και οι διμερεί διαπραγματεύσει. Θα πρέπει να είμαστε ειλικρινεί και να παραδεχτούμε ότι ε, ο δρόμο των πολυμερών συμφωνιών βάσει τη ατζέντα τη Δόχα είναι κάτι που φαίνεται πια δύσκολο. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ρεαλιστέ και γι' αυτό πρώτα απ' όλα να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε όσα προβλέπει ε, η δέσμη μέτρων του Μπαλί. Ε, με την διευκόλυνση των συναλλαγών κυρίω. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε το τέλμα του πολυμερού επίπεδου που έχει επέλθει τα τελευταία χρόνια. Ε, και το να ξαναρχίσουν οι διαπραγματεύσει του γύρω τη Ντόχα χωρί να μην λάβουμε υπόψη τα συμπεράσματα του Μπαλί είναι κάτι που μα φαίνεται εσφαλμένο. Όπως γνωρίζετε υπήρχε προθεσμία της 31ης Ιουλίου για την θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Εμπορικής Διευκόλυνσης, κάτι που δεν το προλάβαμε. Αυτό ελπίζουμε λοιπόν να αλλάξουμε και η Γενική Διεύθυνση Αζεβέντο να μπορέσει να βρει μια θετική λύση στο ερχόμενο διάστημα. Θα θέλαμε για τις υπηρεσίες, για την συμφωνία, για τις για τις ε, ε, υπηρεσίες πληροφορίας και τεχνολογίας, για τα οικολογικά αγαθά, όλες αυτές οι συμφωνίες να ολοκληρωθούν σύντομα. Έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε το σημείο που συναντώνται επιτυχημένα η διμερής προσέγγιση και η πολυμερής προσέγγιση. Να υπογραμμίσουμε εδώ ε, ένα άλλο σημαντικό θέμα, την πρόσβαση στις πρώτες ύλες. Δεν έχουν την ίδια βιομηχανική δομή οι ευρωπαϊκές χώρες. Πολλές επεξεργάζονται απλώς τα αγαθά ή τα υλικά. Εδώ λοιπόν πρέπει να αποφύγουμε τις προστατευτικές τάσεις που έχουν να κάνουν με την αξιόπιστη πρόσβαση και χωρίς στρεβλώσεις της πρώτης ύλη που είναι καθοριστικής σημασίας για την ε, ανταγωνιστικότητα και την παραγωγή. Θα πρέπει λοιπόν οι προτεραιότητες της εμπορικής πολιτικής της Ευρώπης να στηρίζουν ε, την ε, βιομηχανία μας και να αντιμετωπιστούν και οι δεσμολογικοί φραγμοί αλλά όχι μονομερός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εφόσον οι δασμοί που προβλέπουμε εμεί τελικά πλήττουν του παραγωγού μα, προφανώ ακολουθούμε παράδοξη προσέγγιση και γι' αυτό η Προεδρία μα θέλει να αναλάβει συγκεκριμένε πρωτοβουλίε για, να για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Τώρα, για την νομοθετική μας δράση σε θέματα διεθνούς εμπορίου. Η Ιταλική Προεδρία θέλει να ξεπεράσει τα προβλήματα σε δύο άλλα σημαντικά νομοθετήματα τον εξυγχρονισμό των ε, εργαλείων για την εμπορική μας άμυνα, TDI, και το εργαλείο για τους ε, διεθνείς διακονισμούς, IPI. Μας ενδιαφέρει εδώ να μπορούμε να έχουμε συμμετοχή σε δημόσιες προμήθειες τριτών χωρών. Η Επιτροπή ΙΝΤΑ και το Ευρωκοινοβούλιο γενικώ έχουν τοποθετηθεί με σαφή τρόπο θετικά υπέρ αυτών των νομοθετημάτων. Και ήδη στο Συμβούλιο δεν έχουμε δυστυχώ την πλειοψηφία κρατών μελών που θα μπορούσαν να στηρίξουν την πρόοδο ε, των ε, προτάσεων αυτών. Γι' αυτό, με συνεργασία με την Ελληνική Προεδρία, ελπίζουμε ότι θα αναθερμανθεί η συζήτηση στο Συμβούλιο και ελπίζουμε οι συμβιβαστικές μας προτάσεις για τα TDI και τα IPI να γίνουν αποδεκτές. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα για τα εργαλεία αυτά της εμπορικής μας άμυνας θα πρέπει να επιτύχουμε να ισχύσει ο κανόνας του ίσονος δασμού. Εδώ Ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να λάβει υπόψη τι προτάσει μα για κάποιε περιπτώσει σαφών στρεβλώσεων στην αγορά και ελπίζω να μπορέσουμε με ευελιξία να συνεργαστούμε. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορούσε να αποφύγει την έγκριση τεσσάρων εγγράφων εργασιών όπως έχουν ονομαστεί, τι τις γραμμέ, προτού συμφωνήσουν μεταξύ του το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Σε ό,τι αφορά τον κανονισμό για τις διεθνείς προμήθειες, η πρότασή μας, η συμβαστική μας πρόταση έχει ήδη λάβει την θετική άποψη του Κοινοβουλίου. Ελπίζουμε οι ενδιασμοί κάποιων κρατών μελών να ξεπεραστούν με ένα κοινό κείμενο που θα μπορέσει να στηρίξει την κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδίω όταν η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή διαπραγματεύεται τι προποθέσει πρόσβαση ε, των δικών μα κρατών στι δημόσιε προμήθειε τρίτων χωρών. Ελπίζουμε με αυτέ τι νομοθετικέ πρωτοβουλίε να φτάσουμε στο ανάλογο επίπεδο ερήμανση, ώστε να φτάσουμε και σε αίσιο πέρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να ξεπεράσουμε αυτό το αδιέξοδο, ώστε το Συμβούλιο να αποφανθεί και για τα δύο αυτά θέματα που σα ανέφερα από του ερχόμενου μήνε. Τέλο, θα θέλαμε και άλλα ε, νομοθετικά ντοσχέ να προχωρήσουν κυρίως ε, ο κανονισμός που απαγορεύει την εμπορία εργαλείων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της θανατικής ποινής ή για βασανιστήρια ή για ιδιαίτερα σοβαρές, απάνθρωπες ή πίνες. Εδώ θα πρέπει να αποφύγουμε τέτοιου είδου συναλλαγές και την ε, έμεση στήριξη της Ευρώπης τέτοιου είδους ε, φαινομένων. Άλλωστε θα πρέπει να αποφύγουμε και την διακριτική μεταχείριση εις βάρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ για την προσοχή που μου δώσατε και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε επικοδημητικά για να έχουμε έναν ειλικρινή και πολύ συγκεκριμένο διάλογο γι' αυτό, ε, θα ήθελα και το Συμβούλιο όσο το δυνατόν συντομότερα να ξεκινήσει μια εντατική συζήτηση για τη μελλοντική εμπορική μας πολιτική, προκειμένου και η νέα Επιτροπή να, δημοσιεύσει ένα ε, πρόγραμμα με προτεραιότητες για τη νέα της θητεία. Το να έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση αρμοδιότητες για την εμπορική μας πολιτική είναι ένα μεγάλο κατόρθωμα για, τη, για το κοινό μας οικοδόμημα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει από τι δημόσιες διαβουλεύσεις και τον διάλογο των θεσμικών οργάνων που άμεσα έχουν εκλεγεί από τους πολίτες να ε, χαθεί αυτού του είδους η συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι με μεγάλη σαφήνεια παρουσιάσατε τις προτεραιότητες της Τελικής Προεδρίας και νομίζω ότι σε πολλά σημεία αγγίζετε τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να ανοίξω τον πρώτο γύρο απαντήσεων από πλευρά των πολιτικών ομάδων, ακολουθώντα τη σειρά των πολιτικών ομάδων ανάλογα με την ισχύ τη κάθε ομάδο. Στη συνέχεια να δώσω τη δυνατότητα στον Υπουργό να απαντήσει και θα ήθελα να το πω ευθύ εξ αρχή ότι θα επιθυμούσα οι συνάδελφοι να δείξουν μια αυτοπιθαρχία και να μην μιλήσουν πάνω από δύο λεπτά σε ό,τι αφορά τι ερωτήσει που θα θέσουν. Από το ΕΛΚΑ, ο κύριο Κασπάρη. Αξιότιμη κύριε Υπουργέ, σα ευχαριστώ που βρίσκετε σήμερα μαζί μα ε, το πρωί. Θα ήθελα να υπογραμμίσω από πλευρά τη ομάδα μου όλα τα σημεία τα οποία αναφέρετε και θεωρώ ότι πραγματικά είναι πολύ ευρεία η ημερήσια διάταξη, η ατζέντα τη Προεδρία σα για θέματα εμπορικού ενδιαφέροντο. Έχω και κάποιε ανησυχίε, ωστόσο. Καταρχά, ανησυχώ ότι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα υπάρξει μία ανικανότητα σε ό,τι αφορά την ομοθεσία σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια. Θα θυμάστε το τέλος της προηγούμενης εκλογικής περίοδου στο Κοινοβούλιο που έγινε η συζήτηση για τις οικονομικές επιπτώσεις των, ε, της προστασίας επενδύσεων. Μας πήρε πάρα πολύ χρόνο μέχρι να βρούμε μια συνένεση, ένα συμβιβασμό με το Συμβούλιο. Και τώρα η μεταρρύθμιση των εμπορικών προστατευτικών μέτρων και άλλων μέτρων έχουν πάει πίσω στη, στο Συμβουλίο. Και πολύ ανησυχώ ότι αυτό το θέμα δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα πολλά κράτη-μέλη να προχωρήσουν δηλαδή στην νομοθεσία. Ρωτώ λοιπόν, πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια δυνατότητα αυτές οι διαρκείς ε, καθυστερήσεις να μειωθούν στο Συμβούλιο. Δεύτερη ανησυχία. Διμερείς συμφωνίες. Το Συμβούλιο διαπιστώνει πάντα ότι πρόκειται για μεικτή αρμοδιότητα των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό τι σημαίνει ότι θα πρέπει οι συμφωνίες να επικυρωθούν από όλα τα κοινοβούλια. Και σε ό,τι αφορά τις συμφωνίες με την Κολομβία και το Περού, δύο χρόνια ε, κρατάει αυτή τη διαδικασία επικύρωσης και δεν έχει επικυρωθεί καν από τα μισά κράτη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα λοιπόν να σας ζητήσω να, κάνετε, να ξεκινήσετε μια πρωτοβουλία στο Συμβούλιο προκειμένου να διέπονται αυτές οι εμπορικές συμφωνίες ε, από ευρωπαϊκό δίκαιο και να μην είναι μεικτής αρμοδιότητα στο μέλλον. Και τρίτη ανησυχία. Μιλήσατε για τις συμφωνίες που έχουμε ήδη συνάψει ή που πρόκειται να συνάψουμε πολύ σύντομα, Σιγκαπούρου, Εκβαδόρ, Καναδά, θα μπορούσατε να μας πείτε πώς θα διεξαχθεί η διαδικασία επικύρωσης, γιατί νομίζω ότι και πάλι θα τέθει το θέμα της ε, μετάφρασης ε, από πλευρά του Συμβουλίου, θα υπάρξει κάποια δυνατότητα επιτάχυνσης της όλης διαδικασίας, γιατί θα είναι κρίμα αυτές οι συμφωνίες οι οποίες ε, θα ωφελήσουν τους πολίτες μας, να καθυστερήσουν δύο χρόνια παραπάνω για θέματα ε, μετάφρασης. Ευχαριστώ πολύ στους ελληνικράτες τώρα, ο Μάρτιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου για την πλήρη παρουσίαση των θεμάτων του. Όπως είπε και ο προηγούμενος ομιλητής, συμφωνούμε με πολλά θέματα από αυτά που είπε, ιδίω τα σχόλια για την διαφάνεια που έκανε. Θα είναι πολύ σημαντικά για τις δημόσιες συζητήσεις. Τέσσερις, ε, τέσσερις σύντομα ερωτήματα. Μπαλή. Σωστά αναφέρατε ότι ήταν μία μεγάλη επιτυχία. Η Επιτροπή βέβαια πρέπει να κάνει τις διαπραγματεύσεις τώρα. Και αυτή είναι η υπεύθυνη, αλλά πιστεύω ότι θεωρείται πω η Προεδρία, εσεί δηλαδή μπορείτε να μιλήσετε με χώρε όπω την διέζη για να του ζητήσετε να καταλάβουν τη σοβαρότητα τη κατάσταση και να μην θέσουν σε κίνδυνο ολόκληρο το πακέτο του Μπαλί. Δεύτερον, Σάιτα. Συμφωνώ με την αξιολόγησή σας. Πρόκειται για μια επιτυχία. Όπως γνωρίζετε ωστόσο, υπάρχουν σοβαρά ε, σοβαρέ επιφυλάξει στο κοινό σε ό,τι αφορά τη ε, διαδικασία επίλυσης διαφορών. Η Επιτροπή έχει κάνει αξιολόγηση των διαβουλεύσεων που έχει κάνει με την ISDS. Ξέρω ποια είναι η θέση της Επιτροπής. Δεν αφορούσε ολόκληρο το ISDS, αλλά μόνο ζητήτα. Ωστόσο, μήπως θα έπρεπε να μην προχωρήσει περαιτέρω μέχρι ότου έχουμε το, την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Κάτι άλλο, δεν ξέρω αν το αναφέρετε, δεν νομίζω. Ή δεν το κατάλαβα. Μας πίεσαν στο Κοινοβούλιο να προχωρήσουμε γρήγορα στην, και σωστά στην Συμφωνία Όπλων με τις ΗΠΑ. Και το κάναμε, θέλαμε να υπάρξουν οι 50 υπογραφές για την θέση ισχύ της συμφωνίας. Και αυτό θα γινόταν μόνο αν υπήρχε υπογραφή από πλευράς των κρατών της Ένωσης. Από ό,τι ξέρω, μέχρι τώρα, μόνο 8-9 κράτη έχουν 8-9 ε, κράτη δεν έχουν ακόμα υπογράψει την σύμβαση αυτή του ΟΗΕ και αν την υπογράψουν θα τεθεί σε ισχύ. Οπότε θα ήταν χρήσιμο σε επίπεδο Συμβουλίου να ασκηθεί μια κάποια πίεση στα κράτη αυτά. Ξέρω ότι η Ιταλία την υπέγραψε η χώρα σας δηλαδή, αλλά και άλλα κράτη δεν το έχουν κάνει. Τώρα, στις διαφορές για τα θέματα επενδύσεων, βρισκόμαστε στην ίδια κατάσταση τώρα. Ομόφωνα, χτες συμφωνήσαμε ότι δεν ήταν σωστό η Επιτροπή να απειλήσει εκ των προτέρων με νομοθετικά κείμενα. Ποια είναι η άποψή σας ως Προεδρεύων του Συμβουλίου και Πρόεδρος της Επιτροπής ε, της, του Συμβουλίου σχετικά με το θέμα αυτό. Θα ήταν σκόπιμο νομίζετε να στείλουμε από κοινού μια επιστολή στην Επιτροπή αναφέροντας ότι θεωρούμε πως τούτο είναι εσφάλμα, εσφαλμένο ή συντηρητική. Ευχαριστώ. να ευχαριστήσω τον κύριο Υφυπουργό για την πολύ ανοιχτή παρουσίαση που έκανε. Τρεις παρατηρήσεις, σύντομες. Πρώτον, δώσατε σημαντική έμφαση στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σωστό. Μπορεί να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος στα σχέδιά σας για το πώς θα διευκολύνετε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, της Ένωσης σε εξωτερικές αγορές. Η έκθεση που είχαμε στο προηγούμενο κοινοβούλιο μιλούσε για την ευκολότερη πρόσβαση μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε κάποια χρηματοοικονομικά εργαλεία που θα ενίσχυαν την εξαγωγική ικανότητά τους. Έχετε κάποια συγκεκριμένα σχέδια. Αν ναι, θα ήθελα να ακούσουμε δύο λόγια. Δεύτερον, προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, κάτι που όπω ξέρουμε δημιουργεί πονοκεφάλου ε, από καιρού καιρών ε, ε, με συγκεκριμένε χώρες. Θα μας πείτε δύο λόγια για το θέμα. Τρίτον, ένα συγκεκριμένο ζήτημα η πρόοδο τη διαπραγματεύση για, την εμπορική συμφωνία με το Βιετνάμ. Αν κατάλαβα καλά, είπατε ότι η πρόοδος και η ανάπτυξη στη συμφωνία αυτή εμπορικής συνεργασίας εξαρτάται από τις πολιτικές εξελίξεις, την πολιτική κατάσταση στο Βιετνάμ. Δεν ξέρω αν το κατάλαβα σωστά. Δεν ξέρω πάντως κατά πόσον η πολιτική κατάσταση στο Βιετνάμ θα είναι τέτοια που δεν επιτρέπει να συνεχιστούν επιτυχώς οι διαπραγματεύσεις αυτές. Ε, το χρονοδιάγραμμα αν θυμάμαι καλά, αρχικά έλεγε να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις στο τέλος του έτους, δηλαδή στο τέλος της προεδρίας σας. Τι γίνεται με αυτό. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Σάγκε. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Μεταξύ των πολλών που είπατε, σημείωσα την έμφαση η Ένωση να δουλέψει βάσει των αξιών στον κόσμο να δούμε δηλαδή το εμπόριο και σαν ένα πλαίσιο αξιών, όχι μόνο εμπορικά. Με μεγαλύτερη ηγεσία και φιλοδοξία επιδιώκοντας το κοινό συμφέρον, κάτι σημαντικό στο πλαίσιο του Συμβουλίου ιδίω, όπου μερικές φορές τα ε, εθνικά συμφέροντα μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση με το κοινοτικό ή με το κοινό συμφέρον. Ελπίζω ότι η νέα είπα, το είπατε εκπρόσωπος που ξέρετε καλύτερα φαντάζομαι από πολλούς από εμά, θα διασφαλίσει ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή στην εξωτερική πολιτική συμπεριλαμβανομένη και τη εμπορική, διότι φαίνεται μερικέ φορέ ότι οι δύο πολιτικέ ζουν σε διαφορετικού κόσμου. Συγκεκριμένα, μιλήσατε για την εταιρική σχέση με τη ΣΥΠΑ, την συμφωνία. Ε, θέλουμε στις συζητήσεις για συγκεκριμένα θέματα να υπάρξει πλήρης ε, διαφάνεια. Και νομίζω ότι εδώ τα κράτη-μέλη πρέπει να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο, τόσο ώστε τα στοιχεία και τα γεγονότα, αλλά και η αξιολόγηση του πιθανών επιπτώσεων τη συμφωνία αυτής θα μελετηθούν και θα ε, αξιολογηθούν όχι μόνο στα κράτη-μέλη, αλλά ανακλάδο, αναπεριφέρεια. Θα, ζητ... θα έπρεπε να ζητήσετε λοιπόν από τους συναδέλφους σας να αναλάβουν περισσότερο την ευθύνη της συμφωνίας αυτής. Πρέπει τα γεγονότα σε σχέση με το TTIP να φανούν ξεκάθαρα. Τώρα, η διαπραγματεύση για το για την, τη συμφωνία με τα όπλα. Ποια είναι η άποψή σας για την... θα ολοκληρωθεί κατά πάσα πιθανότητα. Ποιες είναι οι απόψεις σας για τις μελλοντικές εμπορικές σχέσεις με το Ιράν και εν γέννη με τις σχέσεις με το Ιράν δεδομένη της ιστορίας που έχουμε τη χώρα αυτή και την ανάγκη να υπάρχει πιο ανεξάρτητη στρατηγική της Ένωσης όταν έχουμε να επικοινωνήσουμε, να συζητήσουμε με μια χώρα που έχει πολλά προβλήματα αλλά έχουμε και κοινά συμφέροντα. Εξαγωγική έλεγχη, τελευταίο θέμα. Η... Το νομοθετικό κείμενο έχει έχει μείνει σε στασιμότητα για πολύ καιρό, παρότι υπάρχουν σημαντικά παραδείγματα που προέρχονται και από την Ιταλία, όπου διαπιστώνουμε ότι επιχειρήσεις όπως το Hacking Team ή το RISPA εξάγουν τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από δικτάτορες. Ο Assad για παράδειγμα, για να καταπιέζει τους πολίτες τους, αλλά και για να παραβιάζει στρατηγικά συμφέροντα της Ένωσης. Πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ ρεαλιστές με την ταχύτητα που εξελίσσονται οι τεχνολογίες αυτές, ούτω ώστε να αναλαμβάνουμε και στα διοικά συμφέροντα υπόψη μας και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η Ένωση θα πρέπει να φροντίζει, και η Προεδρία θα πρέπει να φροντίζει ότι η Ένωση στις επαφές της ε, λαμβάνει υπόψη αυτή την παράμετρο και θέλει να σκόπιμο να κάνετε μια πίεση στο Συμβούλιο για να προχωρήσουν περισσότερο και ταχύτερα στα θέματα του ελέγχου των εξαγωγών. Για τους πράσινους Δεν τον βλέπω. Α, ναι, εδώ είναι. Εκτός μικροφώνου, κύριο Ζαντό. Πρώτο θέμα. Διατλαντική Συμφωνία. Ανήκω σε εκείνους που κατακρίνουν τις διαπραγματεύσεις αυτές. Συνοψίζοντας, να σας πω ότι δεν, ανήκω σε αυτούς που διανέμουν ψευδείς ε, ιδέες ε, για ιδεολογικούς λόγους και είμαι και βαθιά αντιαμερικανός. Αυτή είναι η εικόνα που έχουν για μένα. Αν θέλουμε όμως να έχουμε μια σοβαρή συζήτηση για τα υπέρ και τα κατά της ενδυνάμει αυτής συμφωνίας, είναι σημαντικό να γίνει μια σοβαρή συζήτηση ορθολογική βάσει συγκεκριμένων δεδομένων για το θέμα αυτό γιατί μεταξύ αυτών που διαδίδουν τις ψευδείς ε, αντιαμερικανικές κομματικές ιδέες, έτσι λέει το κείμενο, άκουσα να είναι ο κύριος Γιούνκερ, πρόεδρος της Κομισιόν, ο οποίος ήταν εξαιρετικά επικριτικός σε ό,τι αφορά το μηχανισμό ISDS. Πολλοί συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο εξέφρασαν επίσης αμφιβολίες, επιφυλάξεις, επικρίσεις, ιδίως για την διάσταση επενδύσεων. Θα παρακολουθήσετε, φαντάζομαι, και κατά τη διάρκεια των ευρωεκλογών, ένα κομμάτι της κοινή γνώμης της Ευρώπης έχει σοβαρές επιφυλάξεις για τη συμφωνία αυτή. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να μπορούμε να συζητήσουμε σοβαρά το θέμα αυτό. Λέτε ψευδείς ιδέες σας. Εγώ για ένα χρόνο άκουγα περίπου την, για ένα χρόνο περίπου άκουγα την Επιτροπή να λέει ότι η Διατλαντική Συμφωνία αν γινόταν δεκτή θα έδινε κέρδη 345 ευρώ σε κάθε νοικοκυριό της Ευρώπης μέχρι το 2027. Μετά ένας Ευρωπαίος ε, Επίτροπος Εμπορίου ε, μας είπε ότι όλο αυτό είναι, δεν λέει τίποτα. Όλη η επικοινωνία δηλαδή της Κομισιόν για να προωθήσει την συμφωνία μας είπε ότι δεν έχει κανένα νόημα. Μας αναφέραν ότι θα δημιουργούσαν τεράστιες, τεράστιο ρυθμό θέσεων εργασία, ενώ όταν το Κοινοβούλιο έκανε την αξιολόγηση, είδε την αξιολόγηση της Επιτροπής, ε, με άλλη έρευνα διαπίστωσε ότι δεν είχε γίνει καμία αξιολόγηση από πλευρά τη Επιτροπή για θέματα απασχόληση. Πρέπει λοιπόν να καταφέρουμε να βγούμε από τη σύγχυση, από τις εσφαλμένες ιδέε και να έχουμε μια σοβαρή συζήτηση. Μιλάτε για διαφάνεια και σωστά. Αν η μεγάλη απόφαση της διαφάνειας από πλευρά Συμβουλίου και Επιτροπή είναι να πάψει να είναι εμπιστευτικό έγγραφο η εντολή που είχε δοθεί πριν από 14-15 μήνες και κυκλοφορούσε ούτως ή άλλως παντού, δεν νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ. Πρέπει να προχωρήσουμε πιο μακριά και με πιο σοβαρό τρόπο. Να μιλήσουμε για τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων. Ποια είναι τα έγγραφα των διαπραγματεύσεων στα οποία έχετε πρόσβαση. Έχετε πρόσβαση εσείς στο γραφείο σας, στη Ρώμη, στα διαπραγματευτικά κείμενα όπως προκύπτουν από τα διάφορα round. Τελευταία παρατήρηση. Όντως χρειαζόμαστε μία μεγάλη σοβαρή συζήτηση. Χάρηκα που προσκλήθηκα στο σεμινάριο που οργανώνεται για την Διατλαντική Συμφωνία. Καλή, καλή ιδέα είναι να τη συζητήσουμε. Κοιτάζοντα τόσο τον κατάλογο των προσκεκλημένων, βλέπω βιομήχανου, εργοδότε, δεν βλέπω συνδικάτα, δεν βλέπω κοινωνία πολιτών, δεν βλέπω κοινοβούλιο. Δεν αμφισβητώ λοιπόν ότι το, το σεμινάριο, ε, το επόμενο σεμινάριο που θα κάνετε στη Ρώμη θα έχει ε, και κοινωνία πολιτών και συνδικαλιστές, αλλά χρειάζεται προσπάθειες. Ο κύριος Σόλτς, σας ευχαριστώ πρόεδρε που δεν με, δεν ξεχάσατε. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ ιδιαίτερος ε, για την εκτενή παρουσίαση των προτεραιοτήτων σας. Ωστόσο, είναι τόσο πολλές αυτές οι προτεραιότητες που πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τους επόμενους 6 μήνες και τι δεν θα μπορέσουμε να εφαρμόσουμε και τι θα κληθούμε να αναβάλουμε για την ε, επόμενη Προεδρία. Τρεις-τέσσερις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Αναφερθήκατε στην εισαγωγή σας στην στρατηγική σε εποχή αλλαγής ε, που παρουσιάστηκε τον Ιούνιο το σχετικό πρόγραμμα και σε ό,τι αφορά και θέματα ε, κλειδί, όπως η απασχόληση. Κοιτώντας τις κυρώσεις, για παράδειγμα, στη Ρωσία, σε συνάρτηση με την οξυμένη κατάσταση που επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και τις ε, σχέσεις με την Ρωσική Ομοσπονδία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, οι οικονομικές και εμπορικές ε, κατά συνέπεια σχέσεις κατά πόσο μπορούν να ασκήσουν πραγματική επιρροή στους τρεις στόχους που έχουμε θέσει, στους τρεις πυλώνες ε, σε ό,τι αφορά το 2014 η ευρωπαϊκή οικονομία υπολογίζει μείωση 20-25% σε ό,τι αφορά το ρωσικό εμπόριο. Αυτό φυσικά θα επηρεάσει και τις θέσεις εργασίας. Σε ό,τι αφορά το εμπόριο με την Ουκρανία έχουμε μείον ε, 32% για το τρέχον έτος. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται το έθεσε και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να γνωμοδοτήσουμε ως Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη Συμφωνία Ελευθερού Εμπορίου με την ε, Ουκρανία επειδή θα πρέπει να περάσει γρήγορα. Πώς λοιπόν το Συμβούλιο σκοπεύει να διασφαλίσει ότι αυτή η στόχοθεσία, αυτή οι στόχοι που τέθησαν τον Ιούνιο θα μπορούν να ισχύουν με αξιόπιστο τρόπο τον Ιανουάριο του 2015. Ή μήπω αυτή η στρατηγική θα αποδυναμώσει περαιτέρω την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, η πολιτική δράση και η στοχοθεσία μας πώς θα συνδυαστούν. Δεύτερο σημείο. Μιλήσατε για το εμπόριο, για τα αγαθά που επηρεάζουν το περιβάλλον, όπου θα υπάρξει καινούριο γύρω στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Θεωρώ ότι είναι καλό να διαβουλευτούμε για τα αποτελέσματα του Μπαλί. Το ερώτημα όμως είναι το εξής. Η Προεδρία του Συμβουλίου πώς θα θέσει με νέο τρόπο τα οριζόντια τέτοια θέματα σε ό,τι αφορά με αυτό που είπατε ότι δεν θέλετε σε μη δασμολογικού φραγμούς. Θεωρώ ότι η πολιτική για το περιβάλλον, για το εμπόριο αποτελούν και οι μη δασμολογικοί φραγμοί αποτελούν ε, όρο βασικό σε ό,τι αφορά τρίτον την στρατηγική για τις πρώτες ύλες. Τι σκοπεύετε συγκεκριμένα να κάνετε. Ευχαριστώ. Η FDD λέει ο πρόεδρος, τελευταία ομιλητές. Ο κύριος Ντάρτμουθ δεν είναι εδώ, ο κύριος Ντάρτμουθ. Ποιος ε, θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Υφυπουργέ. Σας ευχαριστώ για την εφράδειά σας που είναι και πολύ της μόδας το τελευταίο καιρό. Δύο πραγματάκια μόνο να σας ρωτήσω. Υποστηρίζετε ότι η κατάργηση των μη δεσμολογικών φραγμών θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις και δεν θα τις ε, θέσει σε κίνδυνο. Τι εννοείτε συγκεκριμένα. Γιατί βάσει της δικής μου εμπειρίας πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις ήδη από καιρό έχουν κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιβιώσουν απλώς τις ξένες αγορές. Εσείς τι ακριβώς εννοείτε. Υποστηρίζετε ότι οι πολυεθνικές δεν θα ωφεληθούν ε, περισσότερο από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εάν έτσι είναι, γιατί μια ρήτρα για την οποία έγινε τέτοια προσπάθεια για το SDS πέρασε. Και γιατί επιδιώκεται τόσο πολύ η απελευθέρωση, τι διδάγματα είχαμε στο παρελθόν από τις προηγούμενες απελευθερώσεις, τόσες συμφωνίες που επιδιώχθηκαν, τι μας έχει φέρει. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας το αποτέλεσμα και δεν είναι καθόλου θετικό. Δηλαδή, αρκεί να σκεφτούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και αυτά που πέτυχαν με την ε, Συμφωνία Ναύτα. Τι ζουν λοιπόν οι αγορές μας, τι ζουν οι εταιρείε μας και εσύ, τι, εσείς τι ακριβώς ε, προτείνετε για τις εταιρείε μας για να τα πάνε καλά βάσει των ε, σοβαρών αποκλήσεων που υπάρχουν εσωτερικά. Θα ήθελα μια συγκεκριμένη απάντηση, όχι μόνο λόγια. Λόγια τα οποία ήταν πολύ ευχάριστα βέβαια όπως είπα και προηγουμένως. Να. Ξεκινώ από τον πρώτο με Κάσπαρη. Η ικανότητα να νομοθετείς έγκαιρα, πριν το TDI και το EPI, είναι κάτι που με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνο. Και ο λόγος για τον οποίο εμείς, ως Ιταλική Προεδρία, αποφασίσαμε να αναζητήσουμε κάποια συμβιβαστική λύση που θα επιτρέψει την έγκριση των δύο αυτών σημαντικών κειμένων. Εφόσον ωστόσο δεν υπάρχει συμφωνία θέλουμε να προχωρήσουμε επίσημα σε ψηφοφορία. Διότι θεωρούμε πως η... αν υπάρξει πιο ευθυγραμμισμένη ε, διαδικασία έγκριση του Συμβούλου θα είναι καλύτερο. Δηλαδή έχουμε ένα πλαίσιο και ένα χρόνο να βρεθεί συμφωνία. Αν δεν έχουμε συμφωνία στο χρόνο αυτό με ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά και ξαναρχίζουμε. Αυτό επιτρέπει να προχωρήσουμε. Αλλιώ θα ήμασταν συνεχώ σε ακινησία χωρί να ξέρουμε ποια θέση να λάβουμε. Είναι λοιπόν προτεραιότητά μα θέλουμε να την προχωρήσουμε και να τη φέρουμε σε ψηφοφορία το Νοέμβριο. Αν δεν, ακόμα και αν δεν υπάρξει πλειοψηφία, αλλά είναι σημαντικό να ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Μικτή, μικτές αρμοδιότητες είναι ένα άλλο θέμα που βρισκομαστε μικτη ειναι ενα αντιμετωπίζουμε στο Συμβούλιο. Πιστεύω ότι Πρέπει να υπάρξει εξαιρετικά σωστή ισορροπία. Οι συμφωνίες αυτές αυξάνονται και ως προς τη διάσταση και ως προς το στόχο και επηρεάζουν τις χώρες πολύ πιο ευθέως. Είναι λοιπόν σημαντικό να μην υπάρχουν καθυστερήσεις στην εκτέλεση των συμφωνιών, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και σωστή παρακολούθηση του αντικτύπου των συμφωνιών αυτών στις στην κάθε χώρα, συζητώντας το θέμα αυτό στο Συμβούλιο. Βεβαίως αυτό δεν ισχύει για το θέμα των μεταφράσεων. Είναι κάπως ε, σουρεαλιστικό να χρειάζεται να περιμένει κανείς 6-8 μήνες για να μεταφραστεί ένα κείμενο. Και αυτό είναι και κατανόητο και για τους εταίρους μας συχνά. Επ' αυτού λοιπόν νομίζω ότι είναι σωστό να γίνει μια συζήτηση στο Συμβούλιο. Για τον κύριο Μάρτιν. Για τον Πάλι είχατε ρωτήσει. Πώς μπορούμε να προχωρήσουμε, πώς μπορεί να συμβάλλει η Προεδρία για την θετική έκβαση των συζητήσεων στον Παλί. Το πρόβλημα είναι η Ινδία. Και δυστυχώς η νέα κυβέρνηση που περιμένουμε ότι θα είναι περισσότερο υπέρ της απελευθέρωσης, τελικά ήταν κατά της υλοποίησης του πρωτοκόλου. Τι πρέπει να κάνουμε. Νομίζω ότι πρέπει να δράσουμε συνολικά ως Ευρώπη, καθιστώντας σαφές προς όλα τα εμπλεκόμενα κράτη ότι δεν θα υπάρξει πρόοδος σε άλλα κομμάτια της ημερήσιας διάταξης ανάπτυξης της δόχα παρά μόνο αν κλείσουμε το trade facilitation στον Μπαλί. Διότι αυτό που έχω καταλάβει από τι διαπραγματεύσει είναι ότι άμα κλείσει μια συμφωνία δεν μπορεί να την ξανασυζητήσει αν θε να τη χρησιμοποιήσει σε κάτι άλλο. Με κάθε σεβασμό λοιπόν προ την Ινδία, η Προεδρία του Συμβουλίου λέει στο πακέτο αυτό προχωράμε, αλλιώ δεν συζητούμε κανένα άλλο κεφάλαιο τη ατζέντα τη Δόχα, ΣΥΤΑ. το ISDS και το ΣΑΙΤΑ. Να σας πω δύο-τρία πράγματα, πέντε λεπτά. Τα κράτη-μέλη έχουν ήδη συμφωνίες με τρίτες χώρες. Στις συμφωνίες αυτές υπάρχει πάντα μία ρήτρα ISDS. Και πρέπει να σας πω ότι 30% περίπου των περιπτώσεων τα κράτη χρησιμοποιούν αυτή τη ρήτρα στις διμερεί συμφωνίες του. Γι' αυτό όταν δώσαμε την εντολή στην Επιτροπή, δώσαμε εντολή για να διαπραγματευτεί και τη ρήτρα ISDS. Τώρα που ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσει και βρισκόμαστε σε φάση μονογραφής, είναι δύσκολο να αλλάξουμε την άποψή μας και να επανεξετάσουμε τη συμφωνία. Η εντύπωση που έχω είναι ότι αν προχωρήσουμε προς τον, τρόπο, προς την κατεύθυνση αυτή θα πρέπει να ξανανοίξουμε όλα τα κεφάλαια της συμφωνίας και να χάσουμε πολύ χρόνο. Για να σας πω την αλήθεια, το θέμα του ISDS συνδέεται πάρα πολύ με τη ΣΥΠΑ, το ξέρουμε. Και αυτό είναι ο λόγος τον οποίο τώρα βρισκόμαστε στη διαδικασία εντοπισμού του ποια είναι η αντιμετώπιση του κοινού, της κοινή γνώμης. Η στάση μας είναι Ολοκληρώθηκε η Σάιτα. Δεν υπάρχει τρόπος να αλλάξουμε την άποψή μας. Βεβαίως μπορούμε να την εγκρίνουμε ή όχι τη Σάιτα, δεν μπορούμε να ανοίξουμε τις διαπραγματεύση του Σάιτα. Που είναι μια πολύ συντηρητική απόδειξη ότι το εμπορικό επιμελητήριο είναι κατά του, της συμφωνίας αυτής, θεωρώντας ότι δεν είναι θετική Αφετέρου, σε όλα τα θέματα ISDS πρέπει να λάβουμε θέση συνεργαζόμενοι ως Συμβούλιο και Κοινοβούλιο για όλες τις άλλες συμφωνίες. Δηλαδή, ξέρετε, η εμπορική πολιτική είναι διαπραγματεύσεις. Αν θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο που διαπραγματευόμαστε, αυτό θα πρέπει να γίνει ε, λαμβάνοντας υπόψη το πώς το αντιμετωπίσουν η άλλη πλευρά αυτό. Για, το TDI, για τα TDI. Είναι λάθος το ότι δίνει guidelines η Επιτροπή όταν έχουμε νομοθετική διαδικασία, την επιταχύνουμε, προσπαθούμε να βρούμε μια συμβαστική λύση. Συναντήθηκα με τον Επίτροπο χτε και του είπα ότι η άποψή, μου, άποψή μας είναι ότι πρέπει να σταματήσει μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεν βλέπω γιατί υπάρχει αυτή η έντονη στάση να προχωρήσουμε χωρίς να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία με τις κυβερνήσεις. Για την ανάγκη 50 υπογραφών για τη συμφωνία του ΟΗΕ για την ε, ε, απαγόρευση εξαγωγής όπλων. Δεν το ξέρω και επιτρέψτε μου να μην απαντήσω για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τι μπορούμε να κάνουμε. Εγώ μιλούσα για την Ταϊλάνδη καταρχάς, όχι το Βιετνάμ, που εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Έχουμε κάποια ανοιχτά θέματα, πρόσβαση στις κρατικές προμήθειες, τα κλωστοφελουργικά, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί για τα θέματα των κλωστοϊφθοντουργικών και πέραν αυτών βέβαια και κάποια άλλα θέματα. Αυτά για το Βιετνάμ. Η Ταϊλάνδη τώρα. Πολύ σημαντική χώρα. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς εξελιχθεί η πολιτική κατάσταση για να δούμε αν μπορούμε να κλείσουμε ή όχι τις διαπραγματεύσεις σύντομα. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δύο πράγματα υπάρχουν εδώ. Πρώτον, όσο περισσότερο περιλαμβάνεις συμφωνίες εμπορικής διευκόλυνσης που έχουν να κάνουν με διαφάνεια, με απλοποίηση των τελωνιακών και άλλων διαδικασιών. Αυτό είναι κρίσιμη σημασία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι η διευκόλυνση και η διαφάνεια είναι βασικό στοιχείο για την πρόσβαση. Υπάρχει ωστόσο και κάτι καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε, ιδίως για τις νέες συμφωνίες ελεύθερου εμποδίου. Μία πρωτοβουλία που πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να θεσπίσουμε είναι η διαδικασία εκπαίδευση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Κάνουμε το ίδιο στην κάτι παρόμοιο στην Ιταλία και πρέπει να δούμε και κάτι αντίστοιχο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από τη στιγμή που υπάρχει λοιπόν το TTIP του ΣΕΤΑ, της συμφωνίας, ε, δεν αλλάζουν τα πράγματα πάρα πολύ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διανομή, πελάτες. Άρα πρέπει να δούμε πώς θα οργανώσουμε κατάρτιση, ε, μαθήματα κατάρτισης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να καταλάβουν καλύτερα και πλήρως ποια εμπόδια υπάρχουν στην αγορά, ποια είναι τα θέματα που πρέπει να δώσουν, στα οποία πρέπει να δώσουν σημασία. Ε, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η εμπορική μας πολιτική εστιάζει καταρχάς στην, στο, αναγνώριση του γεωγραφικού περιορισμού. Κάτι που είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό, ιδίως με την Κίνα. Είπα άλλωστε ότι έχουμε δύο στάδια. Πρώτον, γεωγραφικό περιορισμό και δεύτερον, ευρύτερη ορισμό του γεωγραφικού περιορισμού για να είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν οι διαδικασίες που επιτρέπουν τον έλεγχο της κατάστασης. Δεύτερον, για το πώς πρέπει να συνδυάζουμε καλύτερα εμπορική και εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα είναι ότι πρέπει να χειριστούμε καλύτερα τη δεύτερη φάση της παγκοσμιοποίησης δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε καλή στρατηγική, καλή εμπορική στρατηγική χωρίς γεωστρατηγικές παραμέτρους. Ε, βέβαια δεν θα τα κάνουμε όλα στην Προεδρία μας γιατί έχουμε φιλόδοξο πρόγραμμα αλλά όχι και τόσο φιλόδοξο. Τώρα, ο αντίκτυπος του TTIP, θέμα που θέσατε και οι δύο. Έχουμε πολλά στοιχεία στο DDIP. Η αξιοπιστία των στοιχείων ποικίλει. Κάποια είναι αξιόπιστα, κάποια όχι. Ποιος ξέρει. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Πρώτον, οι Ηνωμένε Πολιτείε σίγουρα θα είναι τα επόμενα χρόνια μία από τις πιο σημαντικές αγορές. Αύξηση 5% το χρόνο των εισαγωγών από τη ΣΥΠΑ. Αυξάνονται αναπτύσσονται. Δεν μπορούμε να χάσουμε την ευκαιρία αυτή. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό για μας, δεδομένου του ότι κάποιες άλλες πηγές εξαγωγών, κατηγορίες εξαγωγών είναι σε δύσκολη θέση, π.χ. η προσδοσία. Άρα, ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να διευκολύνουμε τις διμερείς ανταλλαγές με τις αγορές αυτές που είναι σε καλύτερη κατάσταση, είναι κάτι που πρέπει να γίνει γρήγορα. Μια άλλη παρατήρηση, η δεύτερη παρατήρηση είναι εξή. Οι Ηνωμένε Πολιτείε θα, θα είναι, είναι πιο ανταγωνιστικοί από την Ευρώπη, το ξέρουμε. Λόγω του κόστου τη ενέργεια και πολλών άλλων λόγων. Αν διατηρήσουμε όλα τα εμπόδια, ε, μη δασμολογικά εμπόδια, δασμοί κλπ. Οι επιχειρήσεις μας μπορεί να έχουν ένα ακόμα λόγο για να φύγουν από την Ευρώπη και να πάνε στη ΣΥΠΑ γιατί θέλουν να έχουν την αγορά και αν υπάρχουν εμπόδια θα πάνε εκεί. Χιλιάδες τομείς επηρεάζονται από μη δοσμολογικά εμπόδια. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε διαφορετικά κριτήρια ως προς την ανεκτικότητα της ληστερίωσης. Που σημαίνει ότι ελέγχεται το ζαμπόν που προέρχεται από την Ιταλία και ε, τα κοντέινερ μπλοκάρονται στη ΣΥΠΑ για μήνες. Έχουμε διαφορετικούς κανόνες στα αυτοκίνητα, στο φωτισμό, σε μια σειρά πραγμάτων. Κάτι που αναφέρατε είναι γιατί είναι χρήσιμο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ένωσης. Γιατί αυτές δεν έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν δύο γραμμές παραγωγής χωριστές για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα τους στην ευρωπαϊκή αγορά και την αμερικανική αγορά. Είναι σαφές γιατί λοιπόν τα μη δασμολογικά εμπόδια είναι τόσο σημαντικά. Για να επανέλθω στο θέμα της κυρίας Σάλκε για το Ιράν. Δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Εκεί είναι που κολλάει η εξωτερική πολιτική με την εμπορική. Νομίζω ότι το Ιράν ήταν πολύ σημαντική χώρα για την Ιταλία, για τις εξαγωγές της Ιταλίας. Ωστόσο, τις κυρώσεις που χρειάστηκε να τις επιβάλλουμε τις ερμηνεύσαμε στενά. Και καλά κάναμε. Διότι εμείς είχαμε πει και για τη Ρωσία το ίδιο λέμε ότι πρώτα είναι η εξωτερική και μετά η εμπορική πολιτική. Έλεγχη εξαγωγών. Πιστεύω ότι πρέπει να το δουλέψουμε περαιτέρω. Αν έχετε τα ονόματα τη εταιρεία που κάνουν πωλήσει ε, από την Ιταλία στον ε, Άσαντ, πείτε το μου έτσι από περιέργεια. Να να αναφερθώ στις δικές σας παρατηρήσεις ε, που δεν απάντησα πλήρως. Εγώ δεν είμαι ικανοποιημένο από το θέμα της πρόσβασης στα έγγραφα και το είπα σαφώς στην παρέμβασή μου. Δεν επιλύεται το θέμα μόνο με τη δημοσιοποίηση της εντολής. Υπάρχει ωστόσο διαφορά μεταξύ του να έχει στο ίντερνετ την εντολή γιατί κάποιος το έβαλε επισήμως και άλλο να το έχεις δημοσιευμένο. Είναι η διαφορά γιατί στο εθνικό πλαίσιο οι συζητήσεις ξεκινούν επίσημα μόνο από την εντολή, όχι από πληροφορίες. Η επισημοποιημένη εντολή είναι το ξεκίνημα του τι είναι και του τι δεν είναι στις διαπραγματεύσεις. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα και κοιτάξτε, εγώ δεν, κα, κατηγορώ όποιον λέει ότι είναι επικίνδυνη η TTIP για ότι είναι αντιαμερικάνους. Ούτε, θα το, ούτε το έκανα ούτε θα το κάνω. Δεν, δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου. Εγώ λέγω ότι υπάρχουν επικρίσεις που είναι υπερβολικές, που είναι αβάσιμες το hormone beef, το, το κρέας με ορμόνες, δεν είναι μέσα στο θέμα. Αυτό είπα, ότι δεν μπορούμε να λέμε ότι θα μας γεμίσουν με κρέας με ορμόνες. Το ίδιο ισχύει σε έναν μεγάλο κλάδο των, ε, του, του φυτογειονομικού τομέα. Δεν θα ανατραπεί ολόκληρη η φυτογειονομική πολιτική από αυτό. Αυτό είναι λάθος. Μετά αναφερθήκατε στο ISDS. Και σας λέω, σωστό, αυτό είναι πραγματικό γεγονός ένα πραγματικό θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και πολλά άλλα ζητήματα μπορούν να συζητηθούν. Η δημοσιοποίηση της εντολής δίνει ένα πλαίσιο και ένα ρητό πλαίσιο και επιτρέπει να μεταφέρουμε στις πρωτεύουσε και όχι στα αναγνωστήρια την καταγραφή δεδομένων και πρακτικών που δεν θα είναι ολοκληρωμένα. Έτσι δεν μπορούμε να ανατρέψουμε, ολόκληρη, δεν μπορεί να δώσουμε και την διαπραγματευτική στρατηγική μας στα χέρια των συνομιλητών που είναι και αντίπαλοι. Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε και προς την κατεύθυνση της δημοσιοποίησης. Δεν σας κατηγορώ γιατί Αμερικάνο, είπα, ποτέ δεν το έκανα. Πιστεύω ότι είναι ένα πολύ λεπτό θέμα, πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά. Αλλά να καταλάβουμε τι είναι σε συζήτηση και τι δεν είναι. Δύο παρατηρήσεις. Ο κύριος Σόλτς είπε πώς συνδέουμε τους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε με την εμπορική πολιτική. Πώς τους συνδέουμε, τους συνδέουμε με την εξή τρόπο. Κοιτάξτε, εμείς τα τελευταία, η Ευρώπη δηλαδή, η Δύση πιο σωστά, έκανε μία προσπάθεια περίπλοκη τα τελευταία χρόνια γιατί επέτρεψε εισάγοντας προϊόντα από χώρες αναπτυσσόμενες μπορούσε να αναπτυχθεί η τοπική βιομηχανία στις χώρες εκείνες. Έγιναν οικονομίες παραγωγής που δημιούργησαν απώλεια θέσεων εργασίας σε εμά και έγιναν οικονομίες κατανάλωσης. Γίνονται οικονομίες κατανάλωσης. Τα νούμερα ποικίλουν, αλλά μπορούμε να δώσουμε, θα έλεγα, αρκετά αξιόπιστα ότι υπάρχουν τα επόμενα 15 χρόνια θα υπάρχουν 800 εκατομμύρια νέοι καταναλωτές. Αυτό είναι θετικό για μας. Εμείς επιτρέψαμε να αναπτυχθούν παραγωγικές οικονομίες, υπέστημεν τις επιπτώσεις, τώρα έχουμε όμως αγορές για τα προϊόντα μας. Θα ήταν παράξενο λοιπόν τη στιγμή που εμείς έχουμε ένα μέρισμα να κερδίσουμε από τις επενδύσεις μας, να αποσυρθούμε. Μάλιστα τη στιγμή που θα έπρεπε να είναι πολύ πιο αποφασιστική η εμπορική μας πολιτική και να πούμε στις χώρες που δεν ανοίγονται ακόμα ότι κοιτάξτε, αν αναπτυχθήκατε, αναπτυχθήκατε χάρη στο ότι εμείς σας δώσαμε πρόσβαση στην αγορά μας. Τώρα εσεί πρέπει να δώσετε πρόσβαση στα δικά μας προϊόντα στι δικέ σας αγορές. Και αν δεν το κάνουν με τον τρόπο που πρέπει, είναι να προχωρήσουμε σε όλο και περισσότερες ε, διμερεί συμφωνίες με τις χώρες που θέλουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Και όπω είπα προηγουμένω μεταξύ του TPP, Trans-Pacific Partnership και TTIP και τις συμφωνίες ε, που κάνουμε με τις χώρες του ΑΣΕΑΝ καλύπτουμε το 60% της αγοράς του κόσμου. Αυτή είναι η δεύτερη φάση παγκοσμιοποίησης. Και θα είναι πολύ δύσκολο να αντιταχθούν οι χώρες που δεν είναι μέσα στη συμφωνία αυτή. Αυτό ισχύει και για το Green Goods και για την, ε, και για την Κίνα. Ο μηχανισμός αυτός που είναι σε τρία επίπεδα απαιτεί μια μεγάλη αποφασιστικότητα από τις χώρες την Ευρώπη και τη ΣΥΠΑ στην συνέχιση της διμερούς απελευθέρωσης των εμπορικών συναλλαγών. Μη δεσμολογική φραγμή, ε, πολυεθνικές, απελευθέρωση και ανισότητες. Προσπάθησα να τα απαντήσω με τις προηγούμενες ε, απαντήσεις μου. Οι αποκλήσεις και οι διαφορές που υπάρχουν δυστυχώς ήταν σφάλμα δικό μας, διότι επιτρέψαμε να γίνουμε οικονομίες που απλώς καλύπτουν ανάγκες και ε, να αντιμετωπίσουμε καταναλωτικές οικονομίες. Είχαμε αποπληθωρισμό το 2012 στο διπλάσιο του συνηθισμένου ποσοστού. Ε, οι εξαγωγές είναι η μόνη δυνατότητα ανάπτυξης που έχουν μείνει στις περισσότερες ε, από τις χώρες μας. Είμαστε οικονομίες υποκατάστασης πλέον. Και το περιθώριο αυτό των εξαγωγών είναι το μόνο περιθώριο ανάπτυξη που μας έχει μείνει. Αν δεν υπάρχει απελευθέρωση λοιπόν, δεν θα έχουμε και περαιτέρω δυνατότητα ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε υπερβεί πλέον το χρονικό όριο και μάλιστα κατά πολύ. Και δυστυχώς θα πρέπει στο σημείο αυτό να κλείσει η συζήτηση. Και σε ό,τι αφορά τις οκτώ συναδέλφου που είχαν ζητήσει το λόγο. Επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε παρά το γεγονός ότι είμαι ε, νέος σε αυτή την Επιτροπή. Ένα θέμα με απασχολεί ιδιαίτερα. Όσοι, όσοι μιλούν από το Συμβούλιο ε, λένε ότι είναι υπέρ της διαφάνειας και θέλουν να δημοσιευτεί η εντολή. Άλλοι ομιλητέ μας λένε ότι ε, το επιχείρημα αυτό που χρησιμοποιούν η δικαιολογία της ε, ομόφωνης ψήφου ε, χρησιμοποιείται υπέρ ή κατά όπως το συμφέρει. Καλό θα ήταν λοιπόν να γράψουμε και να ρωτήσουμε αν είναι υπέρ ή όχι της δημοσίευσης των θεμάτων αυτό ή αν η Προεδρία μπορεί να μας πει σε κάποια άλλη συνεδρίαση ποιες κυβερνήσεις είναι κατά της δημοσίευσης της εντολής διαπραγματικής εντολής. Γιατί κάποιες κυβερνήσεις ενδεχομένως να μην το γνωρίζουν αυτό. Το θέτω λοιπόν ως θέμα είτε να μας πει η Προεδρία δηλαδή του Συμβουλίου ποιοι είναι κατά ή να γράψουμε εμείς τις κυβερνήσεις μας και να ρωτήσουμε ποια είναι η επίσημη θέση. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει έτσι αυτή η κατάσταση. Ε, να το πω ως εξή. Ο λόγος για τον οποίο ζητήσαμε με γραπτή επιστολή τη δημοσίευση της εντολής είναι ακριβώς ο λόγος που αναφέρατε. Με αυτή τη γραπτή επιστολή θα δοθούν και επίσημες απαντήσεις. Το θέμα είναι τόσο πολιτικά ευαίσθητο που δεν είναι σε καμία περίπτωση αποδεκτό να προκύψουν θέσεις και τοποθετήσεις και κλεισμένα των θυρών. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο φρόντισα να συνταχθεί επιστολή και προς του συναδέλφους ώστε τουλάχιστον να μην υπάρχει υποχρέωση, καταναγκασμός δηλαδή, αλλά να δοθούν κάποιες διευκρινήσεις σε σχέση με τα ερωτήματα που δόθηκαν. Μόλις τις έχω θα φροντίσω να ενημερωθείτε. Μάλιστα και έτσι ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτηση με τον κύριο Υπουργό. Σας ευχαριστώ εκ νέου ιδιαίτερως και νομίζω ότι πολλά θέματα ιδιαίτερα σημαντικά τα αναφέρατε, τα εξηγήσατε και επαναλαμβάνω ότι οι θέσεις μας προσεγγίζουν πολύ μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σε πολλά ζητήματα. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσει να συνεχίσει η καλή συνεργασία του επόμενου μήνε, προκειμένου μέχρι τα τέλη του έτου να έχουμε ψηφίσει το TDI και να έχουμε διευκρινίσει πολλά από τα θέματα τα οποία θίξαμε. Σα ευχαριστώ πολύ και σα εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ. Yeah. μας Αγαπητοί συνάδελφοι, να περάσουμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη, συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Και κατά δεύτερον, θα ήθελα να σας πω ότι επειδή έχουμε ξεπεράσει τα όρια τα χρονικά, το 7 θα το αναβάλουμε για το απόγευμα, για την απόγευμα την συνεδρίαση. Ο κύριος Ζάχραντιλ δήλωσε ότι μπορεί να δεχτεί αυτή την αναβολή, άρα να κάτσουμε να συζητήσουμε τον προϋπολογισμό. Το λόγο λοιπόν θα δώσω στον κύριο Μπούγκε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η ερώτησή μου έχει να κάνει και, που έκανα πριν από λίγο στον Υφυπουργό, είχε να κάνει και με τις εμπειρίες που είχα σε ό,τι αφορά τα θέματα προϋπολογισμού, σε ό,τι αφορά δηλαδή την ε, ειδική πλειοψηφία που χρησιμοποιείται συνήθως, αλλά με μια εξαίρεση το θέμα Γαλιλαίο, το οποίο εξακολουθούμε να, εξακολουθεί το Συμβούλιο να χρησιμοποιεί αυτή τη δικαιολογία της ε, ομόφωνης ψήφου. Και θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα κάνουμε με το πολιτικό αυτό θέμα. Σε ό,τι αφορά τις ε, τροπολογίες που κατατίθηκαν και για το ψήφισμα έγιναν 15 τροπολογίες, 4 προτάσεις από πλευρά ε, δικής μας. Προσπάθησα με τις διάφορες ε, ομάδες να καταλήξω στις συμβαστικές προτάσεις. Τις έχω διαβιβάσει για την παράγραφο 1 και 6 να συμπεριλάβω τις ανησυχίες των διαφορών ομάδων σε ό,τι αφορά τα διάφορα αμφιλεγόμενα θέματα, σε ό,τι αφορά τα επιχειρηματικά κέντρα στην Ινδία, την Ταϊλάνδη και αλλού, όπου αναφέρουμε τα θέματα που μας ανησυχούν σε ό,τι αφορά την προστιθέμενη αξία, σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα. Και βάσει λοιπόν των αποτελεσμάτων αυτών θα δούμε πώς θα ασχοληθούμε περαιτέρω με το θέμα αυτό. Επιτρέψτε μου τώρα να πω το εξή για τις τέσσερις ε, αλλαγές ό,τι αφορά τις τροπολογίες που έχουμε προτείνει για τον προϋπολογισμό. Έχουμε μία τροπολογία την οποία κατέθεσα εγώ σε ό,τι αφορά τη συζήτηση της προηγούμενης συνεδρίασης όπου συζητήσαμε το θέμα των απαραίτητων πόρων σε ό,τι αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προπολογισμό δεδομένων του δεδομένου του μεγάλου αριθμού ε, συμφωνίων ελευθερου που διαπραγματεύσεων. Κατά δεύτερον, ε, τροπολογία ΣΑΚΕ σε ό,τι αφορά την στρατηγική επικοινωνία και την αύξηση των μέσων. Εγώ τα εξέτασα το θέμα αυτά, τα θέματα αυτά επισταμένως, αλλά θεωρώ δεδομένως και τη συζήτηση που διεξάγεται στην παρούσα φάση δεν θα καταφέρουμε να θέσουμε αυτό το θέμα και να πούμε ότι θέλουμε τη στρατηγική αυτή επικοινωνία, θέλουμε να διαθέσουμε τους σχετικούς πόρους. Παρ' όλα αυτά, σε ό,τι αφορά την πρόταση του κυρίου Σόλτ, σε ό,τι αφορά τα θέματα τα κατεπήγοντα, με προβληματίζει η διόγκωση των δομών, η μόνιμη διόγκωση των δομών αυτών στα πλαίσια του Κοινοβουλίου χωρίς να υπάρξει προηγουμένω μια σωστή ανάλυση του τι θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε. Γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε ξεφύγει έχουν ξεφύγει οι συνάδελφοι. Άρα τίνω να μην συμφωνήσουν, να σας πω την αλήθεια, με αυτές τις ε, καθεπίγουσες δομές. Σε ό,τι αφορά τις προτάσεις του συναδέλφου Αρένα, θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να μας πει το εξής. Μπορεί να υποστηρίξει τα συμφέροντα αυτά το θέμα είναι ποια κατεπήγοντα έργα θα τύχουν υποστήριξη τελικά. Γιατί πάντα υπάρχει αυτή η συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει αλληλεοεπικάλυψη εργασιών, υπάρχουν έργα τα οποία δύσκολα μπορούν να ολοκληρωθούν. Να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ποια είναι η άποψή της για τα πολιτικά αυτά προγράμματα, τα πολιτικά αυτά έργα. Δεδομένων και όσων συμπεριλαμβάνονται και προβλέπονται ε, από τις ε, δραστηριότητες σταθεροποίησης προκειμένου να τα λάβουμε υπόψη αυτά για το απογευματινό μας θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ο πρόεδρος, ένας ε, συνάδελφος, δύο συνάδελφοι μόνο έχουν ζητήσει το λόγο. Α, ναι, τρεις. Εντάξει, κάτι γίνεται. Βίνκλερ, Μάρτιν, Σόλτς, Κέλλα. Ευχαριστώ, πρόεδρε και ευχαριστώ τον συνάδελφο Μπέγκε για αυτήν την πολύ σημαντική πληροφόρηση. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και να δώσω έμφαση σε κάτι που ανέφερε και ο εισηγητής. Την τροπολογία για τα για τα μεταλλεύματα τα, μάλλον τα μεταλλεύματα των, ε, τα ορυχεία των ε, συγκρούσεων conflict minerals όπως έχουμε δει και οι Ηνωμένε Πολιτείε κάνουν κάποια βήματα για την ρύθμιση του θέματος αυτού με, την, ε, τον νόμο Dodd-Frank και τέτοιους νόμους θα πρέπει να προβλέψει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μπορέσουμε να παρέμβουμε στην πράξη και πιστεύω ότι θα ήταν εφικτό κάτι τέτοιο, Καλό θα ήταν να στηριχθεί η τροπολογία αυτή, αλλά θα πρέπει να ακούσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, θα είμαι πολύ σύντομος. Συμφωνούμε με τον εισηγητή και την πρότασή του για τον προπολογισμό, αλλά δεν μπορούμε να στηρίξουμε την τροπολογία για τα ευρωπαϊκά επιχειρησιακά κέντρα. Επιχειρηματικά μάλλον κέντρα, διότι για τα τέσσερα πιλωτικά προγράμματα, τουλάχιστον και τα τέσσερα μπορούμε να τα στηρίξουμε. Έχουμε ανέκαθεν τα στηρίξει αυτήν την προσέγγιση ως Επιτροπή και αλλού το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Βίνκλερ εν μέρει απήντησε το ερώτημα για τα, για τα μεταλλεύματα των... Ε, από περιοχές με εχθροπραξίες είναι πολύ σημαντικά για συγκεκριμένες χώρες και πρέπει να φροντίσουμε τουλάχιστον εδώ να μην υπάρχει σύγκρουση με τα εργαλεία σταθεροποίησης. Ο Χέλμουτ Σόλτσα, ευχαριστώ πάρα πολύ Μπέρντα. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πρόταση των συμβαστικών λύσεων σε ό,τι αφορά αλλά και για την γνωμοδότηση της Επιτροπής, θα την υποστηρίζουμε, συμφωνούμε με τη γενικότερη κατεύθυνση. Θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που είπε για τα πιλωτικά έργα και την αντίρρηση που είχε για αυτό που προτείναμε εμείς για τα πιλωτικά αυτά έργα. Μετά από τις εξηγήσει του Ιταλού Υφυπουργού εξ ονόματος της Προεδρίας για την εμπορική πολιτική, νομίζω ότι κατέστησε σαφές πως η εμπορική πολιτική διαμορφώνεται από συμβάσεις, από συμφωνίες και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει ε, τον αντίκτυπο της κάθε διμερού συμφωνίας σε όλες τις άλλες συμφωνίες. Άρα, μία απόπειρα θα έπρεπε να γίνει από δικής μας πλευράς να δούμε ποια είναι η δυνατότητα να αύξησης του αντικτύπου αυτού συμπεριλαμβάνοντας όσο πιο πολλούς εμπλεκόμενους φορείς γίνεται. Και νομίζω ότι αυτό θα ήταν προς το συμφέρον το δημοκρατικό. Να μπουν από πλευρά του Κοινοβουλίου οι ανησυχίε του για τα έργα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ η κυρία Κέλλερ. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον εισηγητή για την δουλειά του. Και εμείς στηρίζουμε την πρόθεση αυτή για τα μεταλλεύματα των εχθροπαξιών και θα φροντίσουμε με την έκθεση αυτή νομίζω να τοποθετηθούμε για το θέμα αυτό. Είναι καλό λοιπόν που θα υπάρχουν και σχετικά πιλωτικά προγράμματα. Και για την παρακολούθηση του εμπορίου, Trade Watch, το πιλωτικό αυτό πρόγραμμα το στηρίζουμε. Ήδη έχουμε οργανώσει σεμινάρια και εργαστήρια για τέτοιου είδου πρωτοβουλίε. Νομίζω λοιπόν ότι το να αναλύουμε κάθε φορά που εντοπίζονται τα προβλήματα και τι έχει γίνει ω κάποια χρονική στιγμή είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό ε, διότι αυτό το πρόγραμμα είναι σημαντικό, αλλά οι υπόλοιπε προσεγγίσεις που επιδιώξαμε δεν ήταν πολύ επιτυχημένε γιατί δεν έχει αρκετού πόρου στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι τόσε πολλέ οι εμπορικέ συμφωνίε που είναι αντικείμενο διαπραγματεύσεων ταυτόχρονα και τόσε πολλέ διαρκώ προκύπτουν πέραν τη τακτική νομοθεσία και τη νομοθετική διαδικασία, που πραγματικά υπάρχει έλλειψη πόρων, έλλειψη δυνατοτήτων ε, και εμπειρογνωμοσύνης. Εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και στην Επιτροπή μας έχουμε πολύ εξόλογο προσωπικό αλλά δεν μπορούν να παρακολουθούν τις χιλιάδες σελίδες της κάθε μιας από τις εμπορικές μας ε, συμφωνίες είναι πολύ μεγάλο όγκο, γι' αυτό είναι πολύ καλή ιδέα να προσπαθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ω τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει δώσει ικανοποιητικέ απαντήσει. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτού του είδου την παρακολούθηση και τον έλεγχο θα πρέπει να ασκεί το κοινοβούλιο. Αυτό είναι ο ρόλο μα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να τα καταφέρουμε με όλα αυτά τα τόσο περίπλοκα θέματα και την τόσο ε, κατακαιρματισμένη αυτή η διαχείριση των εμπορικών θυμάτων. Σας ευχαριστούμε πάντως για το σχετικό γνωμοδότηση που υποβάλλατε, διότι είναι πραγματικά σημαντικό την ε, παρακολούθηση των θεμάτων, την ε, προσοχή που τους δίνουμε, να την εντείνουμε και όχι απλώς να προβλέπουμε περισσότερα χρήματα για τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Χρειάζονται συστηματικές συζητήσεις, χρειάζεται προσφορά ειδική γνώσης και κυρίως μια επιβράδυνση, διότι το θέμα είναι η ποιότητα και όχι η ποσότητα. Για αυτόν τον σκοπό λοιπόν και προς αυτήν την κατεύθυνση που βάλουμε τροπολογίες. Ευχαριστούμε και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο, κύριος ο κύριος Διποντέ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Μπέγκε και όλα τα μέλη της Επιτροπής για το έργο τους και το ενδιαφέρον τους τα θέματα αυτά. Πολύ σύντομα να σχολιάσω μερικές από τις τροπολογίες που ακούστηκαν σήμερα το πρωί. Πρώτα απ' όλα για τους ανθρώπινους πόρους. Ευχαριστώ για τη στήριξή σας. Σημειώνω τα όσα υπόθηκαν για την τροπολογία, την ε, απόδοση επιπλέον πόρων. Αυτή τη στιγμή δεν έχω περαιτέρω σχόλια για τη συγκεκριμένη τροπολογία. Σε ό,τι αφορά την τροπολογία για τους εταίρους, σημειώνω το ενδιαφέρον σας για τα κατά πόσον θα πρέπει να έχει μια συνολική στρατηγική ενημέρωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εμπορικές συμφωνίες, ιδίως για τις διαπραγματεύσεις TTIP, έχει εντείνει τις σχετικές προσπάθειες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη με πολύ συγκεκριμένα ενημερωτικά δελτία, με μεταδόσεις στο διαδίκτυο, με συζητήσεις με τους κοινωνικούς εταίρους θα συνεχίσουμε τις σχετικές προσπάθειες και σε αυτόν τον τομέα. Ε, για το πιλωτικό πρόγραμμα TradeBots, παρακολούθηση του βορείου, εδώ απλώς να επαναλάβω κάτι που έχω ξαναπεί στην Επιτροπή σας τον περασμένο Ιούλιο, ότι συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι το πιλωτικό πρόγραμμα TradeBots καλύπτεται από το πρόγραμμα για τις συναντήσεις με την κοινωνία των πολιτών. Εκεί ενημερώνονται οι πρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και γίνονται σχετικές συζητήσεις με, συστηματικές, ε, με συστηματικά ραντεβού όπου οι ενώσεις των πολιτών και ενημερώνονται αλλά και αντιδρούν. Ξέρετε τι έγινε με τη συμβουλευτική ομάδα για τις διαπραγματεύσεις TTIP. Λόγου χάρη έχει δημιουργηθεί τέτοια ομάδα και Νομίζω ότι με τη δημοσίευση ενημερωτικών Φιλανδίων και τη διεξαγωγή δημοσίων διαβουλεύσεων έχουμε κληρώσει τις απαιτήσει για, να, για διαφάνεια. Όσο για τα ορυκτά που είναι πολλές φορές αιτία σειράξεων. εδώ για την περίπτωση του Κονγκόλογου χάρη έχουμε ήδη λάβει μέτρα σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΒΚΟ και υπάρχει και η σχετική τροπολογία την οποία σημειώνουμε. Αλλά για να απαντήσω στο ερώτημά σας, εμείς θεωρούμε ότι διαφορετικά προγράμματα και πρωτοβουλίες ήδη ισχύουν πέραν του προγράμματος για τις νέες ε, δράσεις, συνεργασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα αυτά λαμβάνονται πολύ προσεκτικά υπόψη Ήδη λοιπόν κάποια προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και κάποια από τα προγραμματιζόμενα θα δώσουν καλύτερη απόκριση στα θέματα διαφάνειας και ιδίως για τα ορυκτά που είναι αντικείμενο ανθρωπραξιών όχι μόνο στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αλλά και σε άλλες περιοχές. Κάποια παραδείγματα τέτοιων προγραμμάτων και πρωτοβουλειών που βρίσκονται σε εξέλιξη, εάν τι γίνεται με το Ευρωπαϊκό Εργαλείο για την Σταθερότητα, θα δείτε ότι υπάρχει στήριξη για την εφαρμογή της ε, περιφερειακής πρωτοβουλίας των μεγάλων λιμνών που καλύπτει πόρους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, η καθοδήγηση του ΟΟΣΑ για την στήριξη περιοχών που πλήττονται ιδιαίτερα και περιέχουν ε, και ε, αποτελούν πεδίο ορυκτών που είναι αιτία σειράξεων. Στο Μπουρούντι, στη Ρουάντα, στην Ουγκάντα και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ ε, συνεργάζονται για να μπορέσει η τοπική κοινωνία των πολιτών να βρουν κάποιες ικανοποιητικές λύσεις για ζητήματα όπως η κατανομή των γεών ή των φυσικών πόρων. Ήδη προβλέπεται λοιπόν και γι' αυτό ένα κονδύλι αλλά και μια πρωτοβουλία για την διαφάνεια με διευρυμένο πεδίο ώστε να υπάρχει διαφάνεια για την αλυσίδα προμήθειας και την υπεύθυνη εκμετάλλευση φυσικών πόρων. Άρα ε, το θέμα της διαφάνειας για τα ορυκτά των συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή των μεγάλων λιμνών είναι προγράμματα που ήδη τα έχουμε σκεφτεί και προγραμματίσει, όπως για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Και ευχαρίστως να ενημερώνουμε την Επιτροπή σας συστηματικά για αυτά. Και όσο για τα επιχειρηματικά κέντρα, η θέση μας εδώ είναι γνωστή σας, την έχω αναφέρει και πάλι στο παρελθόν. Δεν υπάρχει νέα πρωτοβουλία στον ορίζοντα. Δεν υπάρχει πρόγραμμα για τη στήριξη των επιχειρηματικών κέντρων. Με τα νέα εργαλεία για τα 2014 και 2015 καλυπτόμεθα. Σημειώνουμε τη δική σας την ε, αξιολόγηση ότι για μελλοντική χρηματοδότηση καλό είναι να ξανααξιολογηθούν τα επιχειρηματικά κέντρα. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους και τις παρατηρήσεις του και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. για τα διάφορα που μας είπαν για τα πλαιτικά έργα. Να κάτσουν οι συνάδελφοι και να κοιτάξουν τι μας παρουσίασε στο σημείο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την ε, αποφυγή τέτοιων ε, αλληλεπικαλύψεων σε ό,τι αφορά τα έργα αυτά. Δεν είμαι κατά των έργων αυτών, αλλά αν υπάρχουν διάφορες δραστηριότητε ε, που αλληλεπικαλύπτονται, εγώ ως άνθρωπος του προϋπολογισμού είμαι αντίθετος σε τέτοια αλληλεπικάλυψη. Και αυτό λοιπόν νομίζω να το έχουμε υπόψη πριν πάμε στην ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, σήμερα το απόγευμα. Θα ψηφίσουμε το σχέδιο. και θα ορίσουμε την άποψή μας, την τοποθέτησή μας για το προϋπολογισμό. Όπως σας είπα, το επόμενο θέμα στην ημερήσια διαταξία έχει να βληθεί για σήμερα το απόγευμα, στις 3 το απόγευμα. Και περνάμε λοιπόν στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης και χαίρομαι ιδιαίτερος που έχουμε μαζί μας τον καινούριο πρεσβευτή των ΕΙΠΑ εδώ στις Βρυξέλλες, τον ορίζω, τον κύριο Γκάχνα. Δεν θέλω να κάνω μεγάλες εισαγωγές, νομίζω ότι είναι σαφές και αυτό ανέκυψε και το ακούσαμε και στη συζήτηση με τον Ιταλό Υφυπουργό ότι έχουμε πολύ βασικές οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για το TTIP αυτά όλα θα πρέπει να δοθούν υπό καινούριο πρίσμα σε ό,τι αφορά και τις διαπραγματεύσεις ε. αυτές. Αυτό που αποτελεί επιθυμία μας σταθερή είναι να υπάρχει το δυνατόν μεγαλύτερη διαφάνεια και να αξιολογηθεί η πρόοδος που θα σημειωθεί μετά τον Νοέμβριο όταν θα έχουμε τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων ICS και όταν το Κογκρέσο στην Αμερική θα έχει ολοκληρώσει τις εκλογές θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί περαιτέρω η προοπτική των διαπραγματεύσεων. Χαίρομαι ιδιαίτερως λοιπόν που ο κύριος Γκάρνερ έχετε στο κοινοβούλιο στις αρχές της θετίας του. Έχετε λόγο. Good morning. Thank you, Mr. Καλημέρα και ευχαριστώ πρόεδρε για την πρόσκλησή σας να μιλήσω ενώπιον της Επιτροπής σας. Είναι η πρώτη παρουσία μου εδώ σε μια Επιτροπή του Κοινοβουλίου. Όταν ήρθα στις Βρυξέλλες το Μάρτιο Ήδη είχατε ξεκινήσει την προεκλογική περίοδο. Χαίρομαι που λειτουργεί πλήρω το Κοινοβούλιο τώρα και ελπίζω να ξεκινήσουμε μια μακρά και καρποφόρα συζήτηση. Είναι σημαντικό ο κρίσιμο ρόλο του Κοινοβουλίου. Η ταχύ επέκταση των εξουσιών του με κάθε νέα ευρωπαϊκή συνθήκη, μεταξύ των οποίων και την Λισαβόνα, πετέλεσε σημαντική συμβολή στην ενίσχυση τη δημοκρατική νομιμοποίηση των θεσμικών οργάνων τη Ένωση. Στην πρώτη μου παρουσία στο, στη Γερουσία υπογράμμισα την επιθυμία μου για τις καλές σχέσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στην πρώτη δε πολιτική ομιλία μου, αμέσως μετά την άφηξή μου, ανέφερε την επιθυμία αυτή ως ένα από τα, μία από τις τέσσερις βασικές προτεραιότητές μου για τα επόμενα τρία χρόνια. That the Parliament Ξέρω ότι το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή σας ιδίως, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση των διαπραγματεύσεων και την επιτυχία των προθεσμίων για το TTIP. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω στο παρελθόν με πολλά μέλη τη επιτροπή σα, την κυρία Ρέντινγκ που ήταν επίτροπο, τον κύριο Ρεν. Ξέρει η κυρία Ρέντινγκ που βλέπω εδώ τώρα ότι η ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ε, για το Safe Harbor και το Data Privacy είναι μεγάλη, ήταν μεγάλη, είναι μεγάλη προτεραιότητα για μένα που θεωρώ τα θέματα προσωπικών δεδομένων πολύ σοβαρά και θέλω να αποκαταστήσω την εμπιστοσύνη στην ροή των πληροφοριών διατλαντικά. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση η αντιπροσωπεία μας εδώ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πρόσφατη απόφαση του κυρίου Χόλντερ να επεκτείνει στους Ευρωπαίους πολίτες τα ίδια δικαιώματα που έχουν οι Αμερικανοί πολίτες για τα θέματα προσωπικών δεδομένων. Επίσης, χαίρομαι που βλέπω εδώ και τη Μάρικη μετά από πολλούς μήνες. Ξέρω και άλλο, και άλλο με το πίσω, ο Γιώσεφ Ζάγερ δεν είναι εδώ σήμερα, αλλά είναι φίλος που ε, τον ξέρω από την εποχή που ήμουνα στη νομική του Κολούμπια ήταν, ήταν τότε που μόλις είχε εκλεγεί βουλευτής στο πρώτο ελεύθερο Ουγγρικό Κοινοβούλιο. Το 83 ήμουνα και στην Κρακοβία στο Γεγελονιακό Πανεπιστημίο και γνώρισα και άλλο συναδελφός εκεί που ήταν ε, όπου δίδασκε ο πατέρας του άνθρωπος που είναι ε, παράδειγμα για όλους μας, γιατί είχε αμφισβητήσει το, τότε αυταρχικό καθεστώς. Είχα εμπλακεί σε θέματα ευρωπαϊκά εδώ και 23 χρόνια, ως δικηγόρος στην αρχή, ως κυβερνητικός ε, ε, υπάλληλος κατόπιν, ως τραπεζίτης, ως επενδυτής, που ζει και δουλεύει στην Ευρώπη. Από την εποχή που είχα σπουδάσει στην Οξφόρδη και το Κολούμπια, νομική και ευρωπαϊκά, και από τότε που είμαι και ΣΓΕΡ στην Επιτροπή, πιστεύω βαθιά στο ευρωπαϊκό εγχείρημα είναι καλό για την Ευρώπη και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, θεωρώ. Όπως πιστεύω στις Ηνωμένε Πολιτείε, έτσι πιστεύω και στην ικανότητα της Ευρώπης να ανταγωνιστεί και να κερδίσει στο διεθνές εμπόριο. Η Ευρώπη πρέπει να πιστέψει στον εαυτό της. Να πω δύο λόγια ιταλικά στους φίλους μας. Η μαμά μου ήταν από τη Βενετία και μεγάλωσα περήφανος για την ταρική κληρονομιά μου. Έζησα στη Ρώμη την εποχή των μολυβδένιων χρόνων και γύρισα συχνά στην Ιταλία για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους. Επίσης έχω σχέσεις και με τη Γαλλία, να πω στους Γάλλους φίλους μου. Πέρασα χρόνο, αρκετά χρόνο στο Παρίσι σε ένα δικηγορικό γραφείο μεικτό γαλλοαμερικανικό και μετά στις Βρυξέλλες στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Λευκού Οίκου είμαι υπεύθυνο για τις σχέσεις με, τις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Γαλλία. Επίσης ξέρω και Ισπανικά, γιατί ο μπαμπάς μου ήταν πρέσβης τον είπα στην Ισπανία και χάρη στην παρουσία μου εκεί γνώρισα και παντρεύτηκα όλες μια Ισπανίδα. Και είχα την ευκαιρία, συνεχίζει τα γερμανικά ο πρέσβευτής το είπα, είχα την ευκαιρία να δουλέψω και στη Γερμανία, στο Μόναχο, στο ράδιο. Και το 1991, το φθινόπωρο, ήμουνα στο νομικό τμήμα της σχετικής υπηρεσίας. Προφανώ η θέση μου εδώ είναι να προστατεύσω τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είμαι και περήφανο Ευρωπαίος. Τη μισή ζωή μου και όλη τη σταδιοδρόμη μου σχεδόν την πέρασα στην Ευρώπη. Ε, όταν τελείωσα το στάζ μου στην ε, Επιτροπή αναρωτήθηκα τι να κάνω, να γυρίσω πίσω ή να μείνω εδώ και κάτι που δεν έχουν κάνει πολλοί δικηγόροι οι Αμερικανοί αποφάσισα να μείνω εδώ γιατί τότε ξεκινούσε η διεύρυνση προς την Ανατολή και ήταν μια ιστορική στιγμή που ήθελα να είμαι εδώ. Το ίδιο, την ίδια ε, το ίδιο αίσθημα ιστορικής ευκαιρίας το αισθάνομαι και σήμερα, χάρη στην λόγω της παράνομης προσάρτησης της Κρυμαίας από τη Ρωσία και τη συνέχιση της επίθεσης της προς την Ουκρανία που δημιουργεί μια ανθρωπιστική κρίση, η σπουδαιότητα τη της περαιτέρω ενοποίησης της Ευρώπης και των στενότερων διατλαντικών σχέσεων είναι σήμερα προφανέστερος από ποτέ. Ο επίγον χαρακτήρας μιας ε, αύξησης των δαπανών στην άμυνα της Ευρώπης και στην ενεργειακή, κοινή ενεργειακή πολιτική τώρα είναι προφανέστερα. Και η διατλαντική εταιρική σχέση γίνεται βαθύτερη σε εποχές κρίσεως όπως σήμερα. Δεν αλλάζει η κατάσταση σήμερα. Το σημαντικό είναι αν θα δράξουμε τις ευκαιρίες αυτές ή όχι. Σε μια εποχή που η Ρωσία δίνει δυνάμεις και εξοπλισμό στους αποσχιστικά κινήματα της Ανατολικής Ουκρανίας, η Ευρώπη θα ήταν ενδειγμένο η Ευρώπη να θέσει τα περιφερειακά ζητήματα όπως ε, το, ε, τα εμπορικά σε κάποια προοπτική. Έχουμε την ευκαιρία να θα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε επιμακρών τα επόμενα χρόνια. Προσβλέπω σε μια ανοιχτή συζήτηση, έναν ειλικρινή διάλογο. Οι πόρτε ε, του, της αντιπροσωπής μου θα ανοιχτεί πάντα στα μέλη της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου. Προφανώ υπάρχουν διαφωνίε, αλλά διαφωνίε θα πρέπει να υπάρχουν για ουσιαστικά, όχι περιφερειακά θέματα που, με τα οποία ασχολούνται τόσο πολύ τα ΜΕΑ. Ελπίζω οι διαφορές να στηρίζονται σε μια ακριβή ερμηνεία των πολιτικών και συμφερόντων μας. Έχουμε μια κοινή ευθύνη προ το, ε, προς το εκλογικό μας σώμα να καθοδηγούμε και να ενημερώνουμε. Το TTIP είναι το πιο ισχυρό μέσο προώθησης θέσεων εργασίας και συνεργασίας στο παγκόσμιο εμπόριο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν δύσκολες τεχνικές λεπτομέρειες, τον χρόνο είναι ωστόσο αναγκαίες. Υπάρχουν πολλές ε, επιτακτικές γεωπολιτικές αιτίες που επιτρέπουν, που επιβάλλουν να κλείσουμε γρήγορα, ούτω ώστε να υπάρξει μια ε, ολοκληρωμένη συμφωνία που θα δώσει τα αποτελέσματα που θέλουμε, ενώ ταυτόχρονα θα παράσχει και τι ισορροπίε. Ο κ. Καλέντα, ο κ. Υπουργό, τον οποίον είδα, πιστεύει ότι πρέπει να εξετάσουμε και μια ενδιάμεση συμφωνία. Εμεί συνεχίζουμε να πιστεύουμε ωστόσο ότι μόνο μια ολοκληρωμένη συμφωνία θα λειτουργήσει. Έχουμε τα επόμενα χρόνια την ευκαιρία να θέσουμε ένα πρότυπο για μελλοντικέ εμπορικέ συμφωνίε που θα αντικατοπτρίζουν την κοινή εικόνα αντίληψή μα για εμπόριο που στηρίζεται σε κανόνε, διάφορου κανόνε και ένα ρυθμιστικό πλαίσιο. Αν αποτύχουμε οι άλλε χώρε που δεν συμμερίζονται τι αξίε και τα πρότυπά μα, των οποίων ωστόσο το βάρο στο διεθνέ εμπόριο αυξάνεται, θα θέσουν αυτά το πλαίσιο. Το TTIP προωθεί τι θέσει εργασία, ιδίω στι μικρομεσαίες επιχειρήσει που είναι ε, η σπονδυλική στήλη των οικονομιών, κάτι που δεν ε, παρακολουθείται πολύ στην Ευρώπη παρά την αργή ανάπτυξη της Ευρώπης. Θα κερδίσουν και οι δύο πλευρές, αλλά πρέπει να σας πω ότι η Ευρώπη χρειάζεται τη συμφωνευτή περισσότερο. Πώς θα παράσχει η Ευρώπη στους νέους της το μέλλον που θέλουν. Πώς θα μπορέσει η Ευρώπη να πληρώσει ε, τις συντάξεις των συνταξιούχων της χωρίς την ανάπτυξη που απαιτείται. Η TTIP δεν είναι λύση στις προκλήσεις που της δημιουργίας θέσεων εργασίας και ανάπτυξης, αλλά είναι το καλύτερο, με το καλύτερο κίνητρο χωρίς οικονομική επιβάρυνση που θα έχει θετικές επιπτώσεις. Οι Ηνωμένε Πολιτείες ε, πιστεύουν στις διαπραγματεύσεις, έχουν φιλοδοξίες για το, για το αποτέλεσμα. Οι ενδιάμεσες εκλογές δεν θα επηρεάσουν ε, την βούλησή μας αυτή. Προφανώς χρειαζόμαστε τη συμφωνία του Κογκρέσου, αλλά η απουσία αυτής της αρχής προώθησης του εμπορίου δεν εμποδίζει τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε να δημιουργηθεί αυτή η αρχή στις ΗΠΑ. Παρά τα πλονεκτήματα που δημιουργεί το TIP δημιουργεί και ένα κύμα επικρίσεων για δευτερεύοντα θέματα που προσπαθεί να δημιουργήσει φόβο στο κοινό. Αυτοί που έχουν επιφυλάξει για τη συμφωνία και που αρνούνται να πιστέψουν τι διαβεβαιώσεις που του παρέχουν και οι δύο πλευρές απαντούν τα εξή. Εμείς βρισκόμαστε σε ακόμα σχετικά αρχικό στάδιο των διαπραγματεύσεων. Μην προδικάζετε το αποτέλεσμα. Περιμένετε μέχρι ότι έχουμε ολοκληρωμένα κείμενα πριν αποφασίσετε. Ένας από τους μύθους που είναι ότι οι διαπραγματεύσεις γίνονται εν και παραβίστο. Ε, αυτό ωστόσο δεν ισχύει. Ο υπεύθυνος των διαπραγματεύσεων από πλευρά του κ. του Ντεγκχούχτ είπε ότι οι διαπραγματεύσεις είναι οι πιο ανοιχτές που υπάρχουν. Εμείς πάμε στο Κογκρέσο και τα λέμε, η Κομισιόν έχετε σε εσά και σα ενημερώνει. Όπω η ίδια επιτροπή σα είπε πριν από λίγο, ε, είναι δύσκολο να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι πρέπει να σας δώσουμε εμείς περισσότερα στοιχεία για τις διαπραγματεύσεις από αυτά που δίνουμε στο Κογκρέσο. Εμείς παρέχουμε στους ορισθέντες ε, εκπροσώπους του Κογκρέσου να κοιτάζουν τα κείμενα. Υπάρχει τεράστια ενημέρωση προς το κοινό εκατοντάδες ε, ενημερωτικά ε, ομιλίες ε, παρέχονται στις επιχειρήσεις και στην κοινωνία των πολιτών πάμπορες πληροφορίες. Εμείς είμαστε υπέρ της διαφάνειας, αλλά πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει και μια εξισορρόπηση με βάση και άλλους στόχους. Όποιος διαπραγματεύεται σύνθετες διεθνείς συμφωνίες, οποιαδήποτε συμφωνία στην πράξη, και εγώ έχω κάνει εκατοντάδες τέτοιες συμφωνίες, γνωρίζει ότι η απόλυτη διαφάνεια με τους δεν επιτρέπει ε, τον έντιμο διάλογο και την λύση. Επίσης, ένας μύθος είναι ότι είναι μια ατζέντα απορρίθμισης. Παρότι και ο πρόεδρος τον είπα και ο πρόεδρο τη Επιτροπή και πολλοί πολιτικοί ηγέτε και διαπραγματευτέ από τι δύο πλευρέ του Ατλαντικού έχουν υπογραμμίσει ότι δεν υπάρχει τίποτα στο TTIP που θα περιορίσει τι δυνατότητε των κυβερνήσεων να ρυθμίζουν προ όφελο του δημοσίου συμφέροντο ή να μειώσουν το επίπεδο προστασία τη υγεία και, του περιβάλλοντο. Η TTIP δεν θα επιχρεώσει τις ε, ευρωπαϊκέ χώρε να ιδιωτικοποιήσει ε, δημόσιες υπηρεσίες ούτε θα αποκλείσει ούτε θα υποχρεώσει τα κράτη να ιδιωτικοποιήσουν τις επιχειρήσεις κοινή ή την υγεία που είναι εκτός των ε, ε ρυθμίσεων του ΓΚΑΤ. Άλλος μύθος είναι ότι τα στάνταρ στη ΣΥΠΑ είναι χαμηλότερα. Αυτό αγνοεί το γεγονός ότι πολλά στάνταρ, πολλά πρότυπα στη ΣΥΠΑ είναι πολύ ψηλότερα από την Ευρώπη και το ότι εκατομμύρια ε, Ευρωπαίοι Επισκέπτε στι Ηνωμένε Πολιτείε τρώνε το φαΐ μα και οδηγούν τα αυτοκίνητά μας. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να προστατεύουμε τους Αμερικανούς πολίτες όπως και εσείς. Δεν υποχρεώνουμε τους πολίτε μα να τρώνε πράγματα που δεν θέλουν. Θέλουμε να ακούσετε τι λένε οι δικές σας αρχές ασφάλειας τροφίμων, δίνοντας στους πολίτες της Ευρώπης τη δυνατότητα επιλογή Και όχι να στρεβλώνετε στοιχεία που ε, παρουσιάζονται από, με επιστημονικά δεδομένα. Τώρα, για το θέμα του ISDS, ε, ξέρετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ε, υπογράψει πάνω από χίλιες τέτοιες συμφωνίες που περιλαμβάνουν όλες οι συμφωνίες επίλυσης διαφορών, ISDS. Εμείς δεν επιδιώκουμε να δώσουμε, αντίθετα από αυτό που λένε στις επιχειρήσεις το δικαίωμα να ζητήσουν αποζημίωση για ε, διαφυγών, θεωρητικό διαφυγών κέρδους, αλλά να υπάρχει μια εξισορρόπηση μεταξύ της ελευθερίας το, της επιχειρηματικότητας και των δικαιωμάτων των κυβερνήσεων. Θέλουμε να πετύχουμε την ισορροπία αυτή και σε δημερές επίπεδο και καλωσορίζουμε τις ε, συζητήσεις που κάνει η Επιτροπή για το θέμα αυτό προσβλέποντας τα επόμενα βήματα. Τελευταία παρατήρηση. Και οι δύο πλευρές πρέπει να δώσουν έμφαση σε ρεαλιστικές θέσεις αν θέλουν να υπάρξει συμφωνία που θα προωθήσει τα συμφέροντα και των πολιτών και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Αυτό μπορεί να γίνει αν σεβόμαστε τα γεγονότα, μένουμε εστιασμένοι στα θέματα τα σημαντικά και έχουμε ανοιχτό μυαλό. Ευχαριστώ. Thanks a lot. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος, κύριε Πρέσβη. Και τώρα να ανοίξουμε τη συζήτηση. Η κυρία Ρέντινγκ είναι η πρώτη που έχει ζητήσει το λόγο. E είναι μέλος του ΕΛΚ και το ΕΛΚ είναι η μεγαλύτερη ομάδα. Σχόλια εκτός μικροφώνου. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρέσβη, που βρίσκεστε εδώ. Με μεγάλο ενδιαφέρον άκουσα το γεγονός ότι ο Γενικός ε, Εισαγγελέας ε, ζητά την έγκριση του Κογκρέσου για να επεκταθούν οι κανόνες του US Privacy Act, του νόμου για την ιδιωτική σφαίρα και στους πολίτες στην ε, Αμερικανούς πολιτές. Ελπίζω να καταφέρει να συμφωνήσει και η Αμερικανική κυβέρνηση. Να επικεντρωθώ σε ένα θέμα μόνο, γιατί έχουμε πολλά ερωτήματα να σας ε, θέσουμε και να συζητήσουμε σε ό,τι αφορά το TTIP και τις σχέσεις μας. Όλοι γνωρίζουμε ότι έχει... δεν υπάρχει ε, αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο πλευρών ένθεν και ένθεν του Ατλαντικού σε ό,τι αφορά παραβιάσεις των Αμερικανικών επιχειρήσεων για τους κανόνες για την ιδιωτική σφαίρα και ό,τι αφορά τη μη συμμόρφωση των κανόνων των διατλαντικών συμφωνιών. Εδώ και μήνες προσπαθούμε λοιπόν να αν οικοδομήσουμε αυτέ τι σχέσει εμπιστοσύνη και ξέρουμε ότι η προστασία προσωπικών δεδομένων αποτελεί τον ελέφαντα το, στο δωμάτιο, στην αίθουσα, δηλαδή το μεγάλο θέμα το οποίο κανεί δεν θίγει αλλά υπάρχει. Έχω τρει συγκεκριμένε ερωτήσει να σα κάνω. Οι Αμερικανοί ομόλογοι αποδέχονται τι 13 συστάσει που έγιναν τον περασμένο Νοέμβριο σε ό,τι αφορά το safe harbor, οι ασφαλή λιμένες έτσι, να είναι ασφαλείς όντως Κατά δεύτερον, οι Αμερικανοί ομόλογοι συμφωνούν να μείνουν τα θέματα προσωπικών δεδομένων εκτός του TTIP προκειμένου να μην καταστεί περαιτέρω δυσχερή η κατάσταση. Και κατά τρίτον, οι Αμερικανοί ομόλογοι συμφωνούν να αποσύρουν τα αιτήματα τα οποία εκδόθηκαν στις 25 Απριλίου του τρέχοντος έτους σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις teaser για την ελεύθερη ροή τέτοιων δεδομένων χωρίς οποιοδήποτε, οποιοδήποτε έλεγχο για την προστασία των ατόμων. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ο Ντέιβιτ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να προσθέσω τα ευχαριστήρια λόγια μου και τα καλωσορίσματά μου προς τον πρέσβη. Έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Μα είπε ο πρέσβη ότι ήταν ε, διαπραγματευτή σε θέματα εμπορικά εδώ και πολύ καιρό. Θα πρέπει να κατανοήσει ότι έχει αλλάξει η κατάσταση σε ό,τι αφορά τι εμπορικέ διαπραγματεύσει. Πριν από 10 χρόνια και εγώ, ξέρετε, πολλά χρόνια ασχολούμαι με το, ασχολούμαι με το εμπόριο και τι διαπραγματεύσει. Πριν από 10 χρόνια λοιπόν ήταν πολύ περιορισμένο το ενδιαφέρον του κοινού και πολύ μικρό ο πολιτικό έλεγχο, αν θέλετε. Έχει αλλάξει η κατάσταση και οι εμπορικέ συμφωνίες παρακολουθούνται πολύ πιο στενά πλέον και πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να συνηθίσει στο γεγονός ότι θα ε, χτενίσουμε τις συμφωνίες και θα κοιτάξουμε τα θέματα ένα προς ένα, γιατί θα πρέπει να μπορούμε να τα δικαιολογήσουμε και στο εκλογικό μας κοινό σε ό,τι αφορά για παράδειγμα την κατάσταση στην Ουκρανία. Ε, τα πράγματα ίσως να είναι λίγο πιο θεαματικά, αλλά στην πράξη οι εμπορικές συμφωνίες κρίνονται στις λεπτομέρειες. Και ό,τι και να λένε οι διάφοροι, πολλοί Ευρωπαίοι θέλουν α, ε, σχέση με την Αμερική, πολλοί ε, έχουν να πούνε διάφορα πράγματα για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, συνδικάτα τα οποία θεωρούν ότι απειλούνται από το TTIP και εξηγούν συγκεκριμένα ε, γιατί θεωρούν ότι απειλούνται. Από την άλλη, μπορεί ενδεχομένω όντω το TTIP να μην επηρεάσει τα εργασιακά δικαιώματα, αλλά θα πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό. Σε ό,τι αφορά τι διαφωνίε για θέματα επενδύσεων, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα συμφωνήσω με τον πρέσβη. Ε, έχουμε χίλιες 400 διμερείς συμφωνίες και υπάρχει ο κίνδυνος να αυξηθούν τα θέματα διαφωνίας και διαμαχών μεταξύ των ε, επενδυτών. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι «Α, κοιτάξτε, υπάρχει ένα στάτους, δεν υπάρχει πρόβλημα». Υπάρχει πρόβλημα επειδή ακριβώς υπάρχουν οι συμφωνίες που υπάρχουν και ισχύουν σήμερα. Και εγώ το έχω ξεκαθαρίσει στο παρελθόν. Θέλω το TTIP. Σύμφωνο με τον πρέσβη ότι θα είναι καλό και για τις δύο οικονομίες. Και το έχω πει και στην Επιτροπή μας και στην Ολομέλεια ότι θα κρίνω το TTIP σε τελική ανάλυση όταν θα διαμορφωθεί οριστικά. Αλλά θεωρώ ότι έχουμε καθήκον να ακούσουμε τις ανησυχίες και των πολιτικών και του κοινού και των μη κυβερνητικών οργανώσεων και να βεβαιωθούμε ότι θα ληφθούν στα σοβαρά υπόψη αυτές οι ανησυχίες. Η αίμα σας ευχαριστούμε και ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας. Τα καλωσορίζουμε και εμείς και όλοι οι συναδέλφοι στους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές. Ιδίως την δέσμευσή σας για τις διαπραγματεύσεις TTIP και ότι θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στους πολίτες μας αυτά που έχουμε ήδη υποσχεθεί και έχουμε δώσει έμφαση σε αυτά. Βεβαίως αυτό που συμβαίνει με τις διαπραγματεύσεις όπως σωστά είπατε συμπεριλαμβάνει πολλές φήμες και μύθους αλλά ήθελα να μου πείτε τι γίνεται ακριβώς στην ε, Washington και τι γίνεται με την ε, Αμερικανική Αρχή για το Εμπόριο που μπορεί να δώσει λύσεις ε, ή να λάβει αποφάσεις για την εμπορική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Ας σκεφτούμε ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές μπορεί οι Ρεπουμπλικανοί να έχουν την πλειοψηφία στο Κογκρέσο. Τι πιστεύετε ότι θα μπορούσε να γίνει τότε. Η κυρία Σάκη. Ευχαριστώ πρέσβη για τις ε, εισαγωγικές σας παρατηρήσεις. Κρίμα που δεν μιλήσατε και Ολλανδικά αλλά ήταν ε, πολύ σημαντικό ότι μας μιλήσατε με ευθύτητα. Είναι και το δικό μας το στυλ αυτό. Χαίρομαι που εκτιμάτε την, ε, ε, το κύρος του σώματός μας και χαιρόμαστε για τη συνεργασία σας με το Κοινοβούλιο. Πρέπει πραγματικά να υπάρχει αμοιβή εμπιστοσύνη στις διατλαντικές σχέσεις και πιστεύω και εγώ ότι η διαφάνεια ήταν μια από τις υποσχέσεις του Προέδρου Ομπάμα. Καλό θα ήταν να υπάρχει και μια σχετική υπενθύμηση από κύριο Εκτιμώ το γεγονός ότι έχετε επικεντρωθεί στην παγκόσμια προσέγγιση που χρειάζεται, αλλά υπάρχουν δράσεις που παγκοσμίω θα πρέπει να βασίζονται στις θεμελιώδεις αξίες μας. Αξίες που ε, έχουν να κάνουν όχι μόνο με τι, τι πιστεύουμε εμείς εδώ στην Ευρώπη, αλλά και με τα θεμελιώδη δικαιώματα και πώς προστατεύονται στον υπόλοιπο κόσμο. Αυτό το περιμένουμε λοιπόν και από τι ΗΠΑ. Νομίζω ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μα και σε αυτή την Επιτροπή και σε ό,τι αφορά την συμφωνία TTIP. Και καλό θα ήταν αυτό θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ολοκληρωθεί η συμφωνία αυτή. Όταν ε, είχαμε ξεκινήσει και όταν είχε προκύψει το θέμα με το σχιστολιθικό αέριο, ξεκίνησε και συζήτηση για το κατά πόσο τα κάψιμά μα είναι τα σωστά και μήπω χρειάζεται κάτι που να είναι πιο οικολογικό. Καλό θα ήταν ε, οι Αμερικανοί να αυξήσουν εδώ και εκείνη το επίπεδο των φιλοδοξιών τους, όπως βλέπουμε να γίνεται και με την ε, αρχή για την πρόθεση του εμπορίου, αλλά και το πώς προσεγγίζουμε κι εμεί τα μέλη του Κογκρέσου. Εκεί, επειδή και εγώ συμμετέχω στην αντιπροσωπεία για τι σχέσει με τις ΗΠΑ, ε, βλέπουμε να υπάρχει πολύ λιγότερο ενδιαφέρον από την πλευρά των μελών του Κογκρέσου να συναντηθούν μαζί μα. Εάν θέλουμε λοιπόν να προχωρήσουν σωστά οι διαπραγματεύσει TTIP, θα πρέπει και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και από τη Γερουσία να υπάρξει περισσότερη συμμετοχή για να μπορέσουν και η κοινωνία των πολιτών και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να ε, προβάλλουν τις δικές τους προτεραιότητες και να οδηγηθεί σε αίσιο πέρα συμφωνία TTIP. Ε, ελπίζω μάλλον να μεταφέρετε και στην από τον όσα μόλις υπόθηκαν. Ο κύριος Ζαντό, ευχαριστώ πρέσβευτα. Έχετε είπατε κι εσείς κάποια γενικά λόγια προς τους Ευρωπαίους στην εισαγωγή σας. Εγώ χθες είδα τη δεύτερη σεζόν του House of Cards, της γνωστής σειράς, και ο πρόεδρος ε, ήταν ο Jeff Hood. Ευχαριστώ την Αμερικανική ε, βιομηχανία που μας ε, ετοίμασε μια τόσο ωραία δημιουργική σειρά. Τώρα, με την πώληση όπλων, τόσων ευρωπαϊκών ε, ε, χωρών στην Ρωσία και με τα γαλλικά Μιστράλ κυρίως Βρίσκεται της Γαλλίας, βλέπετε τι σχέση μπορεί να υπάρχει μεταξύ εμπορικής πολιτικής και της ανασφάλειας που εσείς ε, επισημάνατε στην αρχή της παρέμβασής σας. Για τις διατλαντικές διαπραγματεύσεις, εγώ θα έλεγα περίπου τα ίδια με τον David Μάρτιν ε, των σοσιαλιστών και δημοκρατών, αλλά με τελείω διαφορετικό συμπέρασμα. Με την ίδια επιφύλαξη καταλήγω στο συμπέρασμα ότι σήμερα δεν θα έπρεπε να γίνει διαπραγμάτευση για αυτήν την συμφωνία, Ακόμα και με τις υπερφιλόδοξες αλλά ε, τελείως κατευθυνόμενες προβλέψεις για ανάπτυξη στην Ευρώπη το 2017. Εγώ πιστεύω ότι θα περιμένουμε το 2027 για να έχουμε ανάπτυξη στην Ευρώπη. Και αναφερθήκατε και στη διαφάνεια των διαπραγματεύσεων. Εδώ υπάρχει ένα στοιχείο που με τη γνώση που έχετε των ευρωπαϊκών χωρών θα πρέπει να σας κάνει να είστε λίγο πιο ε, συγκεκριμένος. Δηλαδή, συνειδητοποιείται ότι ο Ιταλός ε, Υφυπουργός ε, ε, του, Εμπορίου που αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου των Υπουργών για το Εμπόριο δεν οργανώνει συζητήσεις παρά μόνο στο γραφείο του. Πώς το εξηγείται αυτό αντιμετωπίζετε λιγάκι σαν προσκόπου του ε, Ευρωπαίου ηθήνοντε και συνήθω αυτή είναι απέτηση τη Αμερικανική πλευρά. Επίση, δεν είπατε ότι η συμφωνία TTIP είναι, λέτε, κορυφαία προτεραιότητα των Αμερικανών σε θέματα εμπορική πολιτική. Μπορεί να είναι και έτσι, αλλά υπάρχουν επιφυλάξει και σε επίπεδο κοινωνία των πολιτών και κογκρέσου στι ΗΠΑ. Θα θέλαμε να ξέρουμε λίγο περισσότερα. Και τελευταία παρατήρηση. Α φανταστούμε ότι η Αμερικανική πλευρά συνεχίζει να λέει ότι οι δημόσιες προμήθειες είναι θέμα του ομοσπονδιακού κράτους. Και εσεί θέλετε τις δημόσιες προμήθειες να τις ε, εκμεταλλευτείτε για να αναπτύξετε την οικονομία σας. Δεν θέλετε όμως να ε, αλλάξετε κάποιες ρυθμίσεις ή κάποιες, ε, κάποιους κανόνες για τις ε, χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε, γιατί θεωρείται ότι σα προστατεύουν από τι οικονομικέ κρίσει. Το είπε λοιπόν και ο Ντέβιτ Μάρτιν από την ευρωπαϊκή πλευρά. Θεωρούμε ότι η αρχή τη προφύλαξη είναι πολύ σημαντική. Δεν είναι η λογική μα ότι όταν ένα επιστημονικό δεδομένο δεν έχει επαληθευτεί 100% τότε πρόκειται για πολιτική σκοπιμότητα ή παραπλάνηση. Άρα, σε ευρωπαϊκό ε, επίπεδο, εάν αρνηθούμε το μηχανισμό ISDS για την επίλυση εμπορικών διαφορών, τι θα γίνει, ποιο θα είναι το μέλλον αυτής της συμφωνίας. Ευχαριστώ ο Χέλμουντ και πριν ξεκινήσετε Χέλμουντ σας ευχαριστώ, ε, σας παρακαλώ επειδή έχω οκτώ άτομα που έχουν ζητήσει τον λόγο θα κλείσω στο σημείο αυτό την ε, κατάλογο των ομιλητών. Ο Χέλμουντ ευχαριστώ πολύ Μπέρντα, σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρέσβη για την ε, συνοπτική παρουσίαση σε ό,τι αφορά και την ευρωπαϊκή τέτοια αντίληψη. Ναι, συμφωνώ σε θέματα διαφάνειας ότι πρόκειται για θέμα κλειδί στις διαπραγματεύσεις. Και γιατί επικρατεί μεγάλος φόβος σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν είναι σαφές το τι αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Γιατί δεν έχει δημοσιευτεί εντολή σχετική. Ευθύ εξ αρχής λοιπόν. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο σφάλμα που έγινε. Όλοι το καταλαβαίνουν όταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης αποτελούν οι οικονομικές σχέσεις, θέμα τα εμπορίου, πρόκειται για θέματα κατανάλωσης και παραγωγής. Αυτό λοιπόν απασχολεί όλους τους πολίτες στα κράτη-μέλη και ίσως γι' αυτό στην Ευρώπη διεξάγεται ένας ευρύτερο διάλογος για το θέμα αυτό πιο ευρύς από ό,τι στη ΣΥΠΑ. Αλλά βλέπω ότι και στη ΣΥΠΑ είναι έντονες συζητήσεις στην κοινωνία για τις διαπραγματεύσεις. Ποιο είναι το επίκεντρο των διαπραγματεύσεων, λοιπόν. Εγώ, ως μέλος της Επιτροπής Εμπορίου του Κοινοβουλίου, έχω δικαίωμα να περάσω στην αίθουσα ανάγνωσης, η οποία δημιουργηθήκε. Και βλέπω ότι παρά τις ε, παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ISDS, το οποίο δεν ε, συνεχίζεται του οποίου οι διαπραγματεύσει δεν συνεχίζονται, γιατί έγιναν σχετικέ διαβουλεύσει και τον Νοέμβριο λάβαμε υπόψη ποια ήταν τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων. Βλέπω λοιπόν παρόλα αυτά ότι παρόλα αυτά συνεχίζονται οι διαπραγματεύσει. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, οι διαπραγματεύσει είναι κάτι που απασχολεί το κοινό. Το πρόβλημα λοιπόν που αντιμετωπίζουμε είναι πώς θα καταφέρουμε ότι αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων να κοινοποιηθεί στον πολίτη που θα επηρεαστεί από τις διαπραγματεύσεις αυτές. Δεύτερη ερώτηση. Συμφωνώ, συμφωνώ απόλυτα με την ερώτηση της κυρία Ρέντινγκ σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Μόνο τα προσωπικά δεδομένα, γιατί αυτά περιλαμβάνονται στην εμπορική γλώσσα μεταξύ των προϊόντων. Μέσω της τηλεόρασης, των ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων επανέρχονται στην ημερήσια διάταξη γιατί τα προσωπικά δεδομένα σήμερα αποτελούν τμήμα σήμερα και της ψηφιακής ατζέντα. Συνεχίζουμε λοιπόν να πραγματεύουμε την ψηφιακή ατζέντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα uh, Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο. Καταρχάς, θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να συγχαρώ τον πρέσβη για την γλαφυρότητα, τη σαφήνεια και τη συνοπτικότητά του. Μακάρι όλοι οι συνάδελφοι να είχαν την ίδια ικανότητα. σε ό,τι αφορά τις απόψεις της Αμερικανικής κυβέρνησης για το ευρωπαϊκό project, το ευρωπαϊκό έργο, είναι γνωστές. Ίσως όμως ο πρέσβης ε, να μου επέτρεπε να ρωτήσω το εξής, να πω το εξής. Οι τοποθετήσει των πρώην επιτρόπων δεν αποτελούν τις μοναδικές ε, τοποθετήσεις που εκπροσωπούνται εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Ευρωπαϊκό Έργο. Και στην Επιτροπή μας και στην αίθουσα αυτή. Εντάχει, για το TTIP, για τη συμφωνία TTIP. Τεράστιο και πολύ αμφιλεγόμενο το θέμα αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο και ιδιαίτερος ε, ε, επικεντρωνόμαστε στο ISDS ε, σε ό,τι αφορά το μηχανισμό επίλυσης διαφωνιών. Μας μιλήσατε για μετρημένες επιφυλάξεις για το ISDS. Στην Αγγλία στο Ηνωμένο Βασίλειο, ζητώ συγγνώμη, και σε άλλες χώρες. <laughs> Ναι, στην Αγγλία και σε άλλες χώρες. Ίσως κάτι λέει αυτό. Με γλώσσα λανθάνουσα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, λοιπόν, υπάρχουν επιφυλάξεις σημαντικές. Εγώ, ξέρετε, έχω την τιμή να έχω την εμπειρία αυτή. Η κυβέρνηση τον είπα, θα μου επιτρέψει να σας πω, ότι θα πρέπει να κάνει πιο πολλά προκειμένου να εξηγήσει το ISDS και για να περάσει. Και τέλος, ο πρέσβης ήταν πολύ σαφής. Απέχουμε παρασάγκας από ένα οριστικό κείμενο και από μια οριστική συμφωνία. Να είσαστε απόλυτα βεβαίως ότι το κόμμα μου θα καθυστερήσει οποιαδήποτε κρίση για το TTIP, για τη συμφωνία TTIP, μέχρι ότου να υπάρξει δημοσιευμένο ρευστικό κείμενο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαλέσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον κύριο Πρέσβη για τα καλά λόγια για τον πατέρα μου. Έχω τρεις ερωτήσεις για το TTIP. Θα ήθελα καταρχάς να σας ρωτήσω για το... τις αμερικανικές ε, δασμολογικές προβλέψεις για αγαθά. Για τα αγαθά. Θα προτιμούσατε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει το επίπεδο των φιλοδοξιών τη. Μέχρι τον Νοέμβριο μπορούμε να περιμένουμε μια πρόταση. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Ως τώρα η δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο για την ενέργεια σκοπεύετε να ανταποκριθείτε και αν ναι πότε. Και τέλος, αναφέρατε την αρχή προώθησης του εμπορίου. Εάν σωστά κατάλαβα, ο πρόεδρος Ομπάμα δεν θα προσπαθήσει να το περάσει από το Κογκρέσο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και εγώ να συγχαρώ τον ε, για την ε, ε, ειλικρινέστατη και σαφέστατη και ακριβέστατη παρουσίασή του για τη συμφωνία TTIP κυρίως. Μερικές σύντομες ερωτήσεις. Χάρηκα που τον άκουσα να αναφέρεται στην προστασία δεδομένων. Εγώ ως εισηγητής γνωρίζω πολύ καλά ότι είχε προκαλέσει πολλούς τριγμούς αυτό στην Ευρώπη και έθεσε μια ερώτηση και η κυρία Ρέντινγκ, που δεν θα, επαναλάβω, ε, δεν θα την επαναλάβω, αλλά θα με ενδιαφέρει η ίδια απάντηση. Ως προς τη διαφάνεια τώρα. Κάποιες φορές η υπερβολική διαφάνεια μπορεί να οδηγήσει σε παρερμηνίες. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε μια θέση όπου κάποιοι ίσως εκ προθέσεως, ίσως πάλι όχι, τοποθετούνται κατά τη συμφωνία αυτή χωρίς να λαμβάνουν υπόψη όλα τα γεγονότα. Υπάρχουν όντως πολλοί μύθοι, πολλή μυθολογία γύρω από το θέμα, πολλές φήμες. Χρειάζονται αξιόπιστες εξηγήσει λοιπόν από τους διαπραγματευτές ώστε να καταλάβει ο κόσμος τι είναι η πραγματικότητα και τι αυτό που αποτελεί μύθευμα. Και το, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα. δεν θα συμπέσει από αμερικανικής πλευράς η επίλυση του ζητήματος των καυσίμων με τη λήξη της Προεδρίας του κ. Ομπάμα. Ευχαριστώ κύριε Πρέσβη. Καταρχάς, συμφωνώ ότι το TTIP έχει πολύ θετικέ επιπτώσεις και για τη ΣΥΠΑ και για την Ευρώπη και για τις επιχειρήσεις. Και θα επιτρέψει την ανάπτυξη και πέραν των συνόρων μα ενώ ταυτόχρονα έχει μεγάλες ε, δυνατότητες βελτίωσης της κατάστασης ενόψη και της παρούσης κρίσεως στην Ευρώπη. Αλλά αυτό θα το πετύχουμε μόνο αν πείσουμε τους πολίτες μας ότι το θέμα του ISDS θα λυθεί αποτελεσματικά. Ζητήσατε οι διαπραγματεύσεις να στηριχθούν σε ρεαλιστικές προσεγγίσεις. Συμφωνώ μαζί σας. Βέβαια, αυτό απαιτεί παραχωρήσει και από τι δύο πλευρέ. Κατηγορήστε την Ευρώπη για προστατευτισμό. Εσεί έχετε όμω το Buy American. Έχετε μια σειρά ρυθμίσεων που εμποδίζουν ε, τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Άρα χρειάζεται και οι δύο πλευρέ του τραντικού να κάνουν προσπάθειε. Είστε έτοιμοι να επανεξετάσετε το γεγονός ότι ορισμένα Ορισμένε αποφάσει που λαμβάνετε στα πλαίσια θεωρητικά τη ε, προστασία τη εθνική ασφάλεια λειτουργούν προστατευτικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ, κύριε Πρέσβη, για την παρουσίασή σα. Δεν θα επανέλθω στο θέμα τη διαφάνεια. Καταλάβατε ότι εδώ το θέμα είναι προτεραιότητα για μα. Θα σα ζητούσε λοιπόν να καταβάλλετε μια προσπάθεια καλύτερη εξήγηση των θεμάτων. Η έλλειψη διαφάνειας δημιουργεί λάθος εντυπώσεις για το ISDS. Δεν θα επανέλθω. Θέλω ωστόσο να εκφράσω σοβαρότητες επιφυλάξεις για το μηχανισμό αυτό. Δύο μικρές ερωτήσεις. Πρώτον, για την εντολή των διαπραγματεύσεων. Ο Μπαράκ Ομπάμα, από ό,τι καταλάβαμε, δεν θα πάρει διαπραγματευτική εντολή. Δεν πήρε και δεν θα πάρει από το Κογκρέσο πριν τον Νοέμβριο τουλάχιστον. Και ίσως και μετά. Τι ξέρετε περί αυτού. Δεύτερο ερώτημα. Οι διαπραγματευτές από τις δύο πλευρές δεν συμφωνούν από ό,τι φαίνεται για τη συμπερίληψη των γεωγραφικών ενδείξεων στη συμφωνία. Και εδώ υπάρχουν προβλήματα. Τι γνωρίζετε περί αυτού. Ευχαριστούμε. Η κυρία Λεπέν. Κύριε Πρέσβη, συγχαρητήρια. Πραγματικά οι γλωσσικές σας ικανότητες ε, μας αφήνουν αποσβολωμένους. Θέλω να μιλήσω για την κατάσταση στο θέμα της διαφάνειας. Είμαι δικηγόρος. Είναι ευκολότερο να επισκεφθείς έναν φυλακισμένο στη φυλακή από το να διαβάσεις ένα κείμενο του TTIP. Εμείς ε, για να το δούμε έπρεπε να αφήσουμε τα κινητά μας, ούτε στυλό δεν μπορούσαμε να είχαμε στα χέρια μας και ε, είχαμε μπροστά μας έναν ωκεανό εγγράφων χωρίς να μπορούμε να καταλάβουμε ε, τι γινόταν. Εγώ θέλω να ξέρω κατά πόσον οι Αμερικανοί βουλευτές έχουν πρόσβαση στην διαπραγματευτική εντολή, αν ενημερώνονται για τις διαπραγματεύσεις με σαφή τρόπο ή αν υπάρχει η ίδια άρνηση της δημοκρατίας και περιφρόνηση του λαού στη ΣΥΠΑ όπως και στην Ευρώπη. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη φορά στη Γεωργία. Οι αμερικανικές ε, επιχειρήσεις στη Γεωργία είναι πιο παραγωγικές υπό μεγάλες από την Ευρώπη. Η νέα συνθήκη καταργεί όλες τις, ε, όλα, όλα τα τέλη ενώ μειώνει τις ποσοστώσεις σε μια σειρά ευαίσθητων τομέων. Ε, η παραγωγή, οι κανόνες παραγωγής στις δύο περιοχές πρέπει να είναι ίδιες ενώ γνωρίζουμε ότι στις ΗΠΑ χρησιμοποιούνται διαδικασίες που οι Ευρωπαίοι, οι Γάλλοι τουλάχιστον αρνούνται να χρησιμοποιήσουν. Λυπάμαι γι' αυτό. Ε, η Ευρωπαϊκή Γεωργία, ιδίω η Γαλλική Γεωργία, ε, κινδυνεύει να υποστεί επιπτώσεις από αυτή τη σύγκρουση με την εντατικοποιημένη Αμερικανική γεωργία. Η ποιότητα δε της γεωργίας θα είναι στο επίπεδο αυτό που οι Γάλλοι και οι πολλοί άλλοι Ευρωπαίοι απαιτούν, ευθυγραμμιζόμενοι στους Αμερικανικούς κανόνες. Ε, γι' αυτό εμείς είμαστε, εμείς είμαστε αντίθετοι με αυτή την ε, άμεση ανταγωνιστικότητα των δύο μορφών γεωργίας. Πιστεύουμε ότι έχουμε το δικαίωμα να είμαστε αυτάρκεις γεωργικά, αλλά και να μπορούμε να επιλέξουμε τι θα φάμε. Αυτό είναι κοινωνικό δικαίωμα. Κύριε Πρέσβη, έχουμε ε, συμφέρον να θέσουμε στους ε, λαούς μας επιλογές κοινωνιών που δεν τους αντιστοιχούν ουδόλως. Μήπως αυτό δι, κινδυνεύει να μας απομακρύνει από αυτούς, ε, να, μας απομακρύνει αντί να μας φέρει πιο κοντά. Η κυρία Ροντρίγκε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους καλωσορίζοντας τον Αμερικανό πρέσβη και καλά έκανε η η Σπανίδα δηλαδή. Και μπράβο σας. Να σας πω ότι και εγώ αναγνωρίζω τις ευκαιρίες που παρέχει η Συμφωνία για τη βελτίωση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και των ευκαιριών. Όχι όμως οποιαδήποτε συμφωνία. Είπατε στην παρέμβασή σας κάτι εύλογο που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Να μην προδικάζουμε τα αποτελέσματα μιας συμφωνίας που είναι ακόμα σε μια φάση ε, διαπραγμάτευση. Σωστό. Αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι υπάρχουν προδεδικασμένα. Και τούτο διότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης και ανεπαρκής πληροφόρηση. Αν θέλουμε λοιπόν να μην υπάρχουν αυτές οι προκαταλήψεις, και πρέπει να έχουμε κατάλληλη ενημέρωση για να διορθώσουμε ό,τι δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Υπάρχουν δύο θέματα που με ανησυχούν και που θα ήθελα να σας ζητήσω να μου διευκρινίσετε. Πρώτον, αναφερθήκατε στο ότι το επίπεδο ενημέρωσης των ε, Αμερικανών βουλευτών πρέπει να είναι παρόμοιο με αυτό που υπάρχει στην Ευρώπη. Το ερώτημα, το θέμα είναι, έχουμε την ίδια, το ίδιο επίπεδο ενημέρωσης, το δεχόμαστε, διότι μέχρι τώρα η Ευρώπη βουλευτές δεν είναι ικανοποιημένοι με το επίπεδο ενημέρωση. Αγνώ τι λένε οι ομολογοί μου στη ΣΥΠΑ, αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεύτερον, θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η άποψή σα για την αντιμετώπιση του ISDS στην ΣΕΤΑ. Όταν είχε έρθει εδώ ο αντιπρόεδρος, ο, υφυπουργός, ο Ιταλός Υφυπουργός ως εκπρόσωπος της το πρωί αναφέρθηκε στο ότι η θέση των ΗΠΑ στη συμφωνία με τον Καναδά για το θέμα αυτό ήταν ανεπαρκής. Θέλω να ξέρω αν αυτό συμβαίνει, γιατί θεωρείται ανεπαρκής, γιατί έχουμε διαφορετικές θέσεις και θα έπρεπε να δούμε πώς μπορούμε να τις προσεγγίσουμε. Ευχαριστώ. Κύριε Πρέσβη, έχετε το λόγο. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. διότι με τις ερωτήσεις που έγιναν ουσιαστικά κάλυψαν όλο το πεδίο οι συνάδελφοί σας των θεμάτων που μας απασχολούν. Πάντως είναι πολύ σημαντική η ερώτηση της κυρίας Ρέντινγκ. Αυτό που είπατε ε, μας αφορά ιδιαίτερως και ασχολούμαι και με τον λιμένα και με το λεγόμενο DDPA, την Συμφωνία για την ε, συνεργασία των αρχών επιβολής. Ε, ασχολούμαι κυρίως με το κείμενο, με το κείμενο και τη σύνταξή του και έχει μεγάλη σημασία. Η δική μου αντίληψη για το πώς ε, προχωρούν οι διαπραγματεύσεις είναι ότι έχουμε φτάσει πολύ κοντά. Εσείς είπατε για 14 συστάσεις από το περσινό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Οι 11, όπως ξέρετε, είχαν εμπορική ε, χρειά και νομίζω ότι έχουμε φτάσει πολύ κοντά στο αποτέλεσμα. Απλώς ε, είναι θέμα συντακτικό, λεκτικό, μέχρι να επιληθούν ε, οι επιλογές, κάποιες επιλογές λεκτικές. Για τις εξαιρέσεις καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλές ευαισθησίες εδώ για να μην χρησιμοποιούνται συνολικά και να υπάρχουν πραγματικά περιορισμένες μόνον ε, εξαιρέσεις. Εσείς κυρία Ρέντινγκ νομίζω αναφερθήκατε σε μία προσέγγιση σφαιρική που να περιγράφει όλες τις εξαιρέσεις που ισχύουν το, ε, τους όρους βάσει των οποίων οι μυστικές υπηρεσίες θα μπορούν να συλλέγουν δεδομένα. Σίγουρα έχουμε καθυστερήσει αρκετά όχι λόγω κακοπιστίας, αλλά λόγω εσωτερικών θεμάτων μας. Έπρεπε να ε, παραδοθεί στο Λευκό Οίκο έκθεση, να λάβει έγκριση και αυτό καθυστέρησε. Ελπίζουμε πάντως ότι θα είμαστε έτοιμοι εγκαίρως και θα απαντήσουμε επί της ουσίας το έτοιμά σας για μια προσέγγιση συνολική για τις δύο τελευταίες συστάσεις. Όσο για την ερώτησή σας για τις ε, εμπορικές υπηρεσίες, πρέπει να παραδεχτώ ότι δεν γνωρίζω την απάντηση. Θα ενημερωθώ και θα σας απαντήσω. Για αυτό που είπε ο κύριος Μάρτιν, ίσως ε, παρενόησα. Εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί σας δεν ισχύουν σήμερα όσα ίσχυαν προ δεκαετίες. Το αίτημα διαφάνειας έχει σαφώς ενταθεί. Γι' αυτό αναφέρθηκα και στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις στο γεγονός ότι είναι διαφανέστερες οι διαπραγματεύσεις σήμερα από την προ Και το αναγνωρίζουμε. Έχουμε αυξήσει το επίπεδο, την ένταση των διαπραγματεύσεων μέχρι τώρα. Έχουμε δημιουργήσει ε, περισσότερες συμβουλευτικές ομάδες και από τις δύο πλευρές και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από τη δική μας ε, είναι σαφές ότι οι διαβουλεύσεις και οι ακροάσεις, οι ενημερωτικές ε, ακροάσεις, συναντέψεις τύπου που έχουμε τώρα είναι περισσότερες από ό,τι ποτέ. Για το ISDS εδώ ίσως και να διαφωνούμε. Διότι ως πρώην δικηγόρος πρέπει να σας πω ότι αυτό το θέμα είναι από τα αγαπημένα μου. πριν από λίγα χρόνια, όταν ελάχιστοι γνώριζαν την ύπαρξη των μηχανισμών επίλυσης εμπορικών διαφορών, ε, εγώ ήμουν ήδη λάτρης του θέματος. Πραγματικά μετά ε, καλό οποιονδήποτε ενδιαφέρεται στο και λίγο για το θέμα αυτό. Ε, κοιτάξτε το έγγραφο που έχουμε δημοσιεύσει μετά από χρόνια επεξεργασίας για το μοντέλο επίλυσης διαφορών. Λόγου χάρη ενδιασμοί εξφράστηκαν για το SDS το μηχανισμό επίλυση εμπορικών διαφορών, γιατί ο μηχανισμός αυτός θα επηρεάζει την κερδοφορία της τη κερδοφορία των επιχειρήσεων. Δεν ισχύει, διότι βάσει του δικού μας μοντέλου, του BIT και άλλων διατάξεων ε, ISDS, δεν μπορεί κανείς να ε, ε, προσάγει κάποιον ε, για τον οποιονδήποτε λόγο. Πρέπει να αποδειχτεί διακριτική μεταχείριση ότι η φραγμή είναι υψηλή. Υπάρχουν ένα σωρό προποθέσει. Το λέω για όσου από εσά είναι επιφυλακτικοί και διαρκώ επιμένουν στι ίδιε υποθέσει. Τη Βάτενφαλ στην Σουηδία, την περίπτωση των τάκουν στον Καναδά, την περίπτωση Φίλιπ Μόρι. Αυτέ οι υποθέσει συζητούνται ξανά και ξανά. Αλλά πραγματικά να σα πω κάτι. Ουδέποτε δεν θυμούνται οι άνθρωποι ότι αυτές είναι υποθέσεις που έχουν απλώς εκκινηθεί οι διαδικασίες τους. Δεν ξέρουμε τι αποφάσεις θα βγουν. Γι' αυτό πραγματικά να περιμένετε και να έχετε υπομονή για να δείτε τι αποφάσεις θα λάβουν τα δυτικά δικαστήρια. Για το μοντέλο BIT των ΗΠΑ πάντως υπάρχει στο μοντέλο μας ε, σχετική διάταξη που αποφεύγει τις περιττές καταγγελίες ή προβλέπει δυνατότητες και κυβέρνηση για λεπτομερή καθοδήγηση και ερμηνεία των υποχρεώσεων που συνήθως ισχύουν. Υπάρχει περιορισμός στη διάρκεια εντός της οποίας μπορούν να υποβάλουν οι επενδυτές αξιώσεις ή για οργανισμούς που δεν ανήκουν στην κοινωνία των πολιτών που μπορούν να υποβάλουν τις δικές τους καταγγελίε. Υπάρχουν πολλά παραπλανητικά σχόλια για το μηχανισμό ISDS. Εγώ σας ε, ε, εγγυώμαι ότι κάθε κυρίαρχος κράτος, κάθε κυρίαρχος κράτος κάθε κυρίαρχο κράτος προστατεύεται από, αυτή την, ε, από αυτές τις διατάξεις σαν ασπίδα. Υπάρχει μέχρι τώρα από την προηγούμενη σύνοδό μας ε, και από τα διαιτητικά δικαστήρια όπως έχουν λειτουργήσει ως τώρα πλήρη αρχεία για τις υποθέσεις που έχουν εκδικαστεί. Είναι ελάχιστοι αυτοί που κέρδισαν κατά κρατών για την περιβαλλοντική προστασία λοιπόν και όσους ανησυχούν γι' αυτό ε, σε, αυτό σε αυτή την αίθουσα. Δεν είναι ένα εργαλείο για να μπορέσουν οι πολυεθνικές να παραβούν τις διατάξεις ε, προστασίας του περιβάλλοντος. Υπάρχουν έξι υποθέσεις που εκκρεμούν στην Ισπανία λόγω χάρη. Υποθέσεις ISDS. Η Ισπανία είχε εγκρίνει νομοθεσία ώστε οι επενδυτές που ασχολούνται με ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια να επενδύσουν στην Ισπανία. Τελικά θα ανακαλέσουν όμως τους νόμους τους για τους δασμούς και οι επενδυτές δεν θα χτίσουν τα εργοστάσια αυτά στην Ισπανία. Εσείς θεωρείτε ε, ότι ήταν λάθος οι επενδυτές να πούν ότι δεν ήταν δίκαιο. Δεν ήταν δίκαιο αναδρομικά να καταργήσετε τα δασμολογικά ωφέλη που μας έφεραν εδώ για να χτίσουμε κάποια εργοστάσια. Έχω λοιπόν συζητήσει πολύ για το SDS και ευχαρίστω με όποιον έχει αμφιβολίες σε, αυτό σε αυτή την αίθουσα να καθίσουμε και να τα συζητήσουμε και δημερός Για το TPA, κάποιος νομίζω το ανέφερε, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και θα συνεχίσουμε τις σχετικές διαπραγματεύσεις. Δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που προχωρούμε παράλληλα σε πολλές εμπορικές συμφωνίες και σχετικές διαπραγματεύσει. Για μας αυτό δεν είναι πρωτότυπο. Απλώς θα πρέπει να με εμπιστευτείτε. Έχω μιλήσει σε πολλούς που έχουν δει την εξέλιξη με εμπορικών συμφωνίων μέσα από το Κογκρέσο ε, και που ηγούνταν φορέων του επιχειρηματικού κόσμου παγκοσμίω και μου λένε ότι θα έχουμε τη σχετική στήριξη στο Κογκρέσο, αρκεί να είναι καλή συμφωνία. Τους πιστεύω Τώρα πότε θα γίνει αυτό δεν μπορώ να το πω. Οπωσδήποτε όμως, ακόμη και σήμερα πιστεύουμε ότι η συμφωνία αυτή μπορεί να επιτευχθεί στο τέλος της επόμενης χρονιάς. Νομίζω επίσης έγινε κάποια αναφορά στο Μιστράλ, εάν κατάλαβα απόλυτα ό,τι είπατε στα γαλλικά. Ξέρω ότι υπάρχουν και άλλες απόψεις πέραν της δικής μας, αλλά και η γαλλική κυβέρνηση, και κυβέρνηση έχει πολύ συγκεκριμένες απόψεις για την πώληση. Το καταλαβαίνουμε. Εάν υπάρξει ακύρωση θα υποβληθούν πρόστιμα. Θα καταβληθούν μάλλον πρόστιμα. Αλλά Δεδομένων των όσων συμβαίνουν παγκοσμίω, ήταν ευτυχή η συγκυρία για αυτή την πώληση. Λέτε ότι οι προβλέψει για την ανάπτυξη από τη συμφωνία TTIP είναι υπερφιλόδοξε. Μπορεί και να είναι, αλλά μπορεί και όχι. Η απάντησή μου όμω προ εσά είναι ε, και. Τι έγινε. Η Ευρώπη χρειάζεται ανάπτυξη, χρειάζεται δουλειέ. Το μόνο για το που είμαστε βέβαιοι είναι ότι αυτή η συμφωνία και δουλειέ θα φέρει και θα δημιουργήσει ανάπτυξη. Είμαστε πλέον σε, φάση να λέμε ότι, σε θέση να λέμε ότι 0,5% ανάπτυξη είναι πολύ λίγο. Χρειαζόμαστε οποιαδήποτε μονάδα, οποιαδήποτε εκατοστιαία μονάδα ανάπτυξης μπορούμε να αποσπάσουμε σήμερα. Οτιδήποτε μπορεί να μας φέρει δουλειές και ανάπτυξη. Η ψηφιακή ατζέντα, ε, η απελευθέρωση της αγοράς αλλά η συμφωνία TTIP νομίζω ότι πραγματικά θα είναι μια σημαντικότατη κινητήριο δύναμη για την ανάπτυξη, για τη διαφάνεια. Ακούω και παρατηρώ ότι όντω τα περισσότερα σχόλια που έγιναν στέκονται σε αυτό. Ήδη όμω έχω απαντήσει στον κύριο Μάρτιν. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε περισσότερα για τις διαπραγματεύσεις αυτές. Όχι περισσότερα από ό,τι λέμε και στα μέλη του Κογκρέσου. Οι περισσότεροι είναι ικανοποιημένοι με το επίπεδο διαφάνειας. Ε, έχουν πρόσβαση και το προσωπικό ε, που δουλεύει στο Κογκρέσο έχει πρόσβαση στα σχετικά κείμενα. Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερο, δεν μπορούμε να ε, δείξουμε μεγαλύτερη ανταπόκριση στις ανησυχίες που εξέφρασε το Κοινοβούλιο. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Απλώς να προσθέσω. Να είστε βέβαιοι ώστε έχετε επιφυλάξει για τη διαφάνεια. Πηγαίνετε στους ιστοτόπους πριν κρίνετε. Και εκεί να πείτε ότι δεν είμαστε διαφανείς. Υπάρχει τεράστια ποσότητα πληροφοριών. Η διαπραγματευτική εντολή που την αναφέρατε συμπεριλαμβάνεται στον ιστότοπο, ε, ε, στην σελίδα για την ε, ομάδα εργασία του, τη σχετική ομάδα εργασία του Κογκρέσου. Δεν υπάρχει τίποτε το επιβλαβέ στον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τι πληροφορίε. Μπορείτε να ξέρετε τα πάντα σε σχέση με το τι επιδιώκουμε. Για τι δημόσιε προμήθειε και εδώ υπάρχει μια σχετική μυθολογία στι ΗΠΑ. Ναι, ισχύει το Buy American, αλλά ο βαθμός απελευθέρωσης στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ είναι περίπου ε, παρόμοιος. 320 δις είναι το ποσό που ε, καταβάλλεται ε, ετησίως για ομοσπονδιακές και πολιτιακές προμήθειες. Αυτό που ζητάμε από τους Ευρωπαίους είναι απλώς να είναι συγκεκριμένοι για το πού έχουν τα περισσότερα εμπορικά τους συμφέροντα, πού θα έχουν τι σοβαρότερε απαιτήσει. Εκεί θα πρέπει να καθίσουμε και να συζητήσουμε αν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Ναι, είμαστε οι Ηνωμένε Πολιτείε. ξέρετε ποιο είναι το σύστημά μας βάσει του συντάγματος, ότι το ομοσπονδιακό κράτος μπορεί να ε, ορίσει στις πολιτείες ε, πώς θα δαπανίσουν τα κονδύλια τους. Αλλά μπορούμε και να διαπραγματευτούμε μαζί τους το πώς ε, δηλαδή θα πιστεί ένας κυβερνήτης ή ένας νομοθέτης σε επίπεδο πολιτείας ε, να αλλάξει κάποια πράγματα είναι θέμα του τι θα του προτείνουμε για, τις, για τους δασμούς επί των προϊόντων. Η θέση μας παραμένει ίδια. Έχουν υποβληθεί προτάσεις όπως ξέρετε. Θεωρήθηκαν ε, πολύ χαμηλές. Ναι, ενέφετε κι εσείς. Αλλά δεν έχει κλείσει η συζήτηση. Εμείς θα θέλαμε να υπάρχει πλήρης κατάργηση των ε, δασμολογικών φραγμών για τα προϊόντα και τα καθά. Ο Επίτροπο ρώτησε πότε θα βελτιώσουμε την ε, προσφορά μα. Θα γίνει αυτό, αλλά απλώ δεν μπορούμε να σα πούμε ακριβώ πότε. Τώρα για το κεφάλαιο τη ενέργεια. θα δούμε εάν είναι απαραίτητο το κεφάλαιο αυτό, μήπω η ενέργεια μπορεί να καλύπτεται μέσω άλλων κεφαλαίων. Πάντω, ε, καλά κάνετε και το θέτετε το ερώτημα, είναι πολύ σημαντικό, ιδίω επειδή θα έχετε ε, υποψιάζομαι κατά νου τι εξαγωγέ φυσικού αερίου. Δεδομένου του γεωπολιτικού σκηνικού είναι σημαντικό. και ε, το Υπουργείο Ενέργειας έχει υπολογίσει ότι ε, υπάρχει μεγάλη ε, ποσότητα σε κυβικά μέτρα αερίου που εξάγεται. Σημειώνω πάντως ότι το Υπουργείο για την Ενέργεια είναι σημαντικό το ρόλο του εδώ. Δηλαδή, είναι υπογραφή συμφωνία TTIP και ζητήσουμε περισσότερες εξαγωγικέ άδειε αερίου προ την Ευρώπη, νομίζω ότι θα έχουμε αυτομάτως αντική απάντηση. Για το αέριο One Tank όπως έχει ονομαστεί και αυτή την προσέγγιση νομίζω το σχολίασα Και τώρα για την ε, πνευματική ιδιοκτησία έχουμε διαφορετικό σύστημα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στις ΗΠΑ. Αυτό όμω δεν εμπόδισε του εξαγωγεί τροφίμων από την Ευρώπη να λάβουν ένα μεγάλο μερίδιο τη αγορά στι ΗΠΑ. Ξέρετε ότι έχετε ένα πλεόνασμα 6 δι ε, δολαρίων ε, ω Ευρωπαϊκή παραγωγή στι ΗΠΑ. Και είναι γεγονό αυτό το ότι προστατεύουμε με το σύστημα των σημάτων, των εμπορικών μα σημάτων και των γεωγραφικών ενδείξεων κάποια προϊόντα δεν υπήρξε εμπόδιο στο να αυξηθούν οι εξαγωγές από την Ευρώπη. Θεωρούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι Ευρωπαίοι έχουν υπερβάλλει στις ε, απαιτήσεις τους για τις γεωγραφικές ενδείξεις, διότι υπάρχουν ε, κάποιες περιπτώσεις που ε, τα προϊόντα θεωρούμε ότι δεν καλύπτονται από γεωγραφική ένδειξη, αλλά από κάποια πολύ γενός, γενικόλογη αναφορά, όπως η παρμεζάνα λόγου χάρη. Για μας είναι σχεδόν ε, γενική κατηγορία προϊόντος. Δεν αποτελεί ένα, μια γεωγραφική ένδειξη. Τέθηκε τώρα και ένα ερώτημα με τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τα μεγάλα εργοστάσια των ΗΠΑ που είναι ε, μεγάλα εργοστάσια, μα δεν είναι όλες οι αμερικανικές ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις τεράστιες εργοστάσια που θα καταπιούν την Ευρώπη. Έχουμε και εμείς μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις και μικρομεσαίου μεγέθους αγροκτήματα. Σας διαβεβαιώ ότι οι Αμερικανοί καταναλωτές γίνονται όλο και πιο απαιτητικοί. Υπάρχει περιθώριο στην αγορά μας για κάθε είδου προϊόντα και για τα φθηνά και για τα χαμηλότερε ποιότητε ποιότητα, αλλά και για τα υψηλότερη ποιότητα και τα ακριβότερα, ακόμη και τα πλέον ακριβά προϊόντα που μπορεί να εισάγονται από την Ευρώπη. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι μύθο Είναι μύθος ότι η Ευρώπη δεν θα μπορεί να ανταγωνιστεί του Αμερικανούς, αλλά και ότι οι Αμερικανοί δεν θέλουν τα υψηλής σε ευρωπαϊκά προϊόντα, επειδή φτιάχνονται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο και με πολύ συγκεκριμένα συστατικά. Συμφωνώ είναι επιλογή των καταναλωτών. Τι θα ή θα τρώνε τελικά, ποια είναι τα τρόφιμά τους. Αλλά μην αποφασίζουν οι πολιτικοί με, με βάση πολιτικά... πολιτικές Οι... οι Ευρωπαίοι πολλές φορές ψηφίζουν κατά των επιστημονικών συμβουλών ε, ε, της ΕΦΣΑ. Εγώ θα ήθελα οι χώρες που διαφωνούν με την ΕΦΣΑ να δώσουν επιστημονικά στοιχεία και να πούν γιατί διαφωνούν με την Ευρωπαϊκή Αρχή Προστασίας των Τροφίμων. Γιατί διαφωνούν με, τους εθνικούς, με τις Εθνικές Ομοσπονδίες Προστασίας των Τροφίμων. Εκεί θα πρέπει να δούμε τι πρόβλημα έχουμε σήμερα. Και υπήρξε και ένα ερώτημα για τον Μηχανισμό Επίλυση Εμπορικών Διαφορών και την Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία. Δεν έχω δει όλε τι σχετικέ διατάξει τη συμφωνία αυτή ω τώρα και δεν μπορώ να απαντήσω δυστυχώ σήμερα. Πρόεδρε, σα ευχαριστώ που με δεχτήκατε σήμερα και την ευκαιρία να συζητήσουμε τα θέματα αυτά ε, για πολλού μήνε. Θα, θα την έχουμε και στο μέλλον. Όπω είπα και προηγουμένω, η πόρτα μου είναι διαρκώ ανοιχτή με ειλικρινή και διαφανή διάλογο. Ελπίζω ότι πάντοτε τέτοιον θα έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρέσβη και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε περαιτέρω ευκαιρίες να συζητήσουμε, ίσως και να συζητήσουμε το ISD και τις συνέπειες του για το TTIP. Σας ευχαριστώ και πάλι. Συνάδελφοι, σας παρακαλώ να εξέλθετε ησύχως να μείνουν μόνο οι συντονιστές. Συνεδρίαση συντονιστών και κλεισμένων των θυρών. Να φύγουν όλοι όσοι δεν είναι συντονιστές από την αίθουσα.